Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις για Να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα υιοθετείτε η μεσαιρέταξη καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές, αν δεν υπάρχουν λοιπόν η μερίσια διάταξη υιοθετείται όπως τη λάβατε. Και τώρα θα περάσω σε ανακοινώσει του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα με χαρά ανακοινώνω ότι η κυρία Βερονίκ Ματιέ εξελέγει νέα συντονίστρια του ΕΛΚΑ, ο κύριος Γεώργιος Πανικολάου, αντιπρόεδρος, αντι, ε, αναπληρωτή συγγνώμη συντονιστής ε, του ΕΛΚΑ. Να σας συγχαρώ λοιπόν και τους δύο. Έπειτα Ορισμό ηγητών. Η κυρία Τιτμπάουερ από το ΕΛΚ έχει διοριστεί η για το πακέτο θεωρήσεων για την Αρμενία, περιλαμβάνοντα δύο εκθέσει για την επανειστοχή προσώπων που ε, διαμένουν χωρί έγκριση και διευκόλυνση για την έκδοση θεωρήσεων. Έπειτα περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 20 και 21 Μαρτίου 2012 και 3 Σεπτεμβρίου 2012. Αν δεν υπάρχουν αναστάσεις έως στο τέλος της ευρύνη συνεδρίασης θεωρείται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Τώρα, πρέπει να σας ενημερώσω για κάποια πράγματα σχετικά με τις ενεξελίξει διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι Επετέχθη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση για την πρόταση για τροποποίηση του κώδικα στον Οσέγγεν με εισηγή τον κύριο Παπα-Νικολάου. Στον τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο, όπως γνωρίζετε αυτός ο φάκελος είναι τους πέντε φακέλους που είχαν ε, μπλοκάρει στη διάσκεψη των Προέδρων μετά την διαφωνία που υπήρξε στο Συμβούλιο για το πακέτο Σέγγεν. Άρθατε θέση ψηφοφορία μόνο αν το επιτρέψει η διάσκεψη των Προέδρων. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή να μας παρουσιάσει τα κυρία σημεία αυτής της συμφωνίας. Παρακαλώ κύριε ε, Ευχαριστώ πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Αυτή η έκθεση είναι μεταξύ των πέντε που έχουν μπλοκάρει αυτή τη στιγμή από τη διάσκεψη των Προέδρων για τους ε, γνωστούς λόγους. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του τι έχει συμβεί ως τώρα και περιμένω βεβαίω και τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτό το φάκελο κατά τη διάρκεια τη Πολωνική Προεδρία. Συνεχίσαμε κατά την Δανική Προεδρία και ολοκληρώσαμε κατά την Κυπριακή Προεδρία. Μετά την ψήφο στην Επιτροπή μα τον περασμένο Μάρτι, είχαμε τρει ε, συναντήσει ε, στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου με την Δανική Προεδρία και είχαμε σχεδόν καταλήξει συμφωνία, αλλά μετά υπήρξε η απόφαση της των Προέδρων και περιμένουμε λοιπόν και πάλι από τη δίσκηση των Προέδρων να μας δώσει το πράσινο φως για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ε, τις διαπραγματεύσεις κατά την Κυπριακή Προεδρία. Πριν να ξεκινήσω να σας περιγράφω ποια είναι η συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, να σας ευχαριστώ και πάλι όλους τους κοιόδης. Και Βέμπερ, Νοδόσκου, Ντάνοβα, Μακτάιερ, Μένστερ και τον κύριο Κλέης για τη συνεργασία όπως και τη γραμματεία συγκεκριμένα την κυρία Χέλεμ Κάλε. Πρόκειται για τεχνική τροποποίηση του κανονισμού σαν και μια πολύ λοιπόν τεχνική έκθεση αυτή που έχω αναλάβει. Θα θυμάστε και από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει σε προηγούμενες συναντήσει μας. Κατέστη λοιπόν με βάση αυτή την πρόταση αναγκαίο να λάβουμε υπόψη την ε, νεοϊθετήσα πρόταση κανονισμού που είχε εφηρεθεί το 2006 σας θυμίζω αυτή ήταν η τελευταία νομοθεσία με την οδηγία για τις επιστροφές, την καθίδρυση του Frontex και τη νέα νομοθεσία για τις θεωρήσεις και πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις προτάσεις με τον κανονισμό Σάγκεν, λαμβάνοντας υπόψη ε, και την πρακτική εμπειρία των κρατών μελών όπω τη βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, καθώ και τι αναλύσει που έγιναν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όταν πρωτοξεκινήσαμε λοιπόν τη συζήτηση αυτής της έκθεσης, είχαμε συνολικά περίπου 80 α, τροπολογίες, 50 στο σχέδιο έκθεσης και 31 από συναδέλφους και τέλος το Μάρτι σχεδόν ψηφίσαμε ομοφόνος επιτροπολογιών αυτών. Επαναλαμβάνω τρεις συναντήσεις τριμερούς διαλόγου και μία τελική συνάντηση τον περασμένο μήνα όπου ένα ήταν το ακρεμέ ζήτημα το οποίο επιλύσαμε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Αυτό το πρόβλημα αφορούσε τη δυνατότητα, μάλλον την υποχρέωση αναφοράς για την παρουσία ενός συγκεκριμένου προσώπου στο χώρο Σέγγεν. Μετά ή μάλλον σκοπός ε, αυτής της έκθεσης και των τροπολογιών μας ήταν να βελτιώσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο και να ενισχύσουμε τη συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα, προωθώντας περαιτέρω την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια από τα στοιχεία κλειδιά στα οποία καταλήξουμε συμφωνία είναι τα εξή. Και πάλι θέλω να επαναλάβω, πολλές ε, α, παράγραφοι ε, έπρεπε να τροποποιηθούν μετά τον κανονισμό του 2006. Μία σημαντική αλλαγή στον κανονισμό Σέγγεν είναι ο ορισμός και η εισαγωγή των τρίτων σημείων εισόδου στα σύνορα. Είναι κάτι που να συμφωνήσει τους μέλος να δημιουργήσει με μια τρίτη χώρα, ώστε να αναπτύξει ε, καλύτερη ορατότητα στον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Καταφέραμε να διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα επαρκώς με το Συμβούλιο και να καταλήξουμε μια ισορροπημένη θέση. Οπότε κάθε κράτος μέλος που έχει όμορη, τον... ε, τρίτη χώρα μπορεί να συμφωνήσει κάτι τέτοιο όπω η Πολωνία το έχει κάνει. Να έχει τρίτα σημεία διέλευση στα σύνορα αλλά με συγκεκριμένε διατάξεις που προβλέπουν στον κανονισμό Σέγγεν, δηλαδή με ειδικέ διαδικασίε κανόνες, διαδικασίες που αφορούν τα δικαιώματα των συνοριφυλάκων, κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα και την ε, προστασία των δεδομένων ε, που ε, περνούν μέσα από τα συστήματα τα πληροφορική, τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι κατά του ελέγχου και μετά από τι πολλέ τροπολογίε που περάσαμε, έχουμε τον άρθρο 3α πλέον που μιλάει για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Δηλαδή, όταν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό, θα πρέπει πάντοτε να κινούνται μέσα στα πλαίσια ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού και του διεθνού δικαίου. Ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο υπολογισμό τη διαμονή ε, των υπηκότερων κρατών που εισέρχονται στο Σέγγεν. Μια καλύτερη διευκρίνηση του υπολογισμού και συλλογή δεδομένων ε, το, σχετικά με τα πρόσωπα του αρνούνται την είσοδο ε, δεδομένα στατιστικά που πλέον θα πρέπει να αναφέρονται ετησίως στην Eurostat. Επίσης, το κείμενο της Frontex συμπεριλαμβάνεται και αφορά ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για τους συνοριοφύλακες. Δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν. Επίσης, ε, οι διατάξεις για τους ελέγχους στα πλοία είναι καλύτερες πλέον. Θεωρώ σημαντικές προσθήκες στον κανονισμό. Με αυτές τις τεχνικές τροποποιήσεις μπορούμε να πούμε ότι πλέον επικαιροποιεί το κανονισμό Σέγγεν και υπάρχουν και άλλε λεπτομέρειες που μπορώ να σας αναφέρω, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να καταχραστώ του χρόνου σας. Είμαι όμως στη διάθεσή σας, αν το επιθυμείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει λοιπόν συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Δυστυχώ όμω δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να περιμένουμε τη δίσκεψη των Προέδρων να μα επιτρέψει να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με το φάκελο τη κυρία Βέμπερ και τι προτίθεται να κάνει ε, η Ιρλανδική Προεδρία, πώς θα ηγηθεί ε, των διαπραγματεύσεων. Έχουμε έρθει σε επαφές με τους κοιόδε, τους οποίους ευχαριστώ εκ νέου για να συζητήσουμε, να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το τι μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε. Γιατί αν ξεμπλοκαριστεί ο δικό μου φάκελο, ο φάκελο κ. Χωμάγερ, ο οποίο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και είναι αναμονή, να περάσει και αυτό. Πάντως, αν γίνει κάτι τέτοιο και αν ζητήσουμε από τον πρόεδρο τη Επιτροπή να προβεί μια πρωτοβουλία, δηλαδή να απευθύνει μια επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων, για παράδειγμα, το σημαντικό είναι να φανεί καλή συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα και πώς η θέση του Κοινοβουλίου παραμένει ξεκάθαρη και ο ρόλος του Κοινοβουλίου διασφαλίζεται ε, σε ό,τι αφορά τις πραγματεύσεις και παραμένει ο ίδιος ως σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι. Μεγάλη εμπειρία για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που κατέληξα σε μια τέτοια συμφωνία στην Διάλογο. Ήταν μια πραγματική εμπειρία που είχε αίσιο πέρα. Προ το παρόν τουλάχιστον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου. Τώρα η περιγραφή του προγράμματος Δάστης. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 17 Δεκεμβρίου, ο δεύτερος στις 17 και θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή κύριο Κλέης για να μας περιγράψει τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Κύριε Κλέης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό Justice εξετάζεται ταυτόχρονα από την Επιτροπή ΕΛΕΦ, ΛΙΜΠΕ δηλαδή και την Επιτροπή Ζουρί Νόμ Ήδη έγιναν δύο τριμερείς διάλογοι 15 και 17 Δεκεμβρίου και εκεί καταλήξαμε σε μία συμφωνία σε τρία σημεία. Πρώτον, καθορισμός των γενικών στόχων του προγράμματος, τη αιτήση του Κοινοβουλίου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της αμοιβαία αναγνώρισης και αμοιβαία εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαστικών συστημάτων. Δεύτερον, καθορισμό συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος συμφωνήθηκε να τονιστεί ιδιαίτερα το θέμα της επιμόρφωσης του δικαστικού προσωπικού, ιδιαίτερα γλωσσικής και ορολογίας καθώς και τονίστηκε επίσης η σημασία της διαμεθοριακής συνεργασίας χάρη στην πληροφορική. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ήττα δικαιοσύνη και την ήττα μάθηση πάλι μέσω της πληροφορικής ώστε η συνεργασία και η επικοινωνία σε νομικό και δικαστικό επίπεδο να γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερο και να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη. Στις μελλοντικέ διαπραγματεύσει με την Κομισιόν και το Συμβούλιο άλλα σημεία θα εξεταστούν και συζητηθούν, δηλαδή το κατά πόσον, το πώς μάλλον θα ορίσουμε τα προσόντα που πρέπει να έχει το προσωπικό του δικαστικού τομέα το Κοινοβούλιο θα ήθελε να συμπεριληφθεί και το άρθρο 21 της Χάρτας των Θεμελιωδών, ενώ τα άλλα όργανα προτιμούν δικό τους κατάλογο χωριστό. Τώρα για τον καθορισμό των οργάνων που μπορούν να έχουν επιχορηγήσεις, ιδιαίτερα οργανισμών που έχουν μορφή επιχείρησης, Υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που τονίστηκε στις τροπολογίες, δηλαδή το αν όσοι ωφελούνται από το πρόγραμμα θα μπορούν να αναφέρονται στο νομοθετικό τμήμα του κειμένου. Πολλοί τάχθηκαν υπέρ, αλλά με βάση τις εκθέσεις που ενέκριναν οι δύο επιτροπές μας, εμείς θα θέλαμε να εκτιμήσουμε μεν την εξαιρετική δουλειά που έγινε μέχρι τώρα από τις οργανισμούς και υπηρεσίες που υποφελούνται από το πρόγραμμα Justice, αλλά παράλληλα θα θέλαμε η υποβολή αιτήσεων και η χορήγηση επιχορηγήσεων να γίνεται με αντικειμενικό τρόπο και σωστό και ως νομοθέτες και νομοθέτησες θέλουμε να παραμείνουμε ουδέτεροι ως προς τους αιτητάς και ετητρία. Υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία που πρέπει ακόμη να συζητηθούν, δηλαδή οι δείκτες που θα πρέπει να δείχνουν αν ένα πρόγραμμα έχει πετύχει τους στόχους τους και βέβαια το γνωστό και σύνηθες θέμα του κατά πόσον πρέπει να επιμείνει το Κοινοβούλιο είτε στην κατεξουσιοδότηση πράξη είτε στι εκτελεστικέ πράξει. Εμείς είμαστε υπέρ των κατεξουσιοδότηση για να έχουμε έτσι περισσότερο λόγο μπροστά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή που διαφωνούν. Οι διαπραγματεύσεις πάντως αυτές δεν γίνονται στο επίπεδο του τριμερούς διαλόγου για τον οποίο συζητούμε τώρα, διότι υπάρχουν πολλά παρόμοια θέματα που εξετάζονται παράλληλα και που αφορούν πολλά έτη αναφοράς και τα δημοσιονομικά τους έχουν το ίδιο επίσης πρόβλημα και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει κάποια συμφωνία για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Ελπίζουμε επίσης να γίνει αυτό γρήγορα ώστε να μπορέσει να σταλεί στην Ολομέλεια όσο το δυνατόν συντομότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλάις. Τώρα, αύριο στις 11 αμέσως μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών η εισηγήτρια κυρία Γκόντς δεν είναι σήμερα παρούσα γι' αυτό αύριο θα κάνει τη δήλωση που έπρεπε να κάνει σήμερα και τώρα το επόμενο θημείο έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Βάιλα Πλίτκα Φρέιμπεργκα και τον καθηγητή Κόμπαρ που είναι μέλος της υψηλού επίπεδου ομάδας που ιδρύθηκε για να καταλήξει σε συστάσεις για την προώθηση της ελευθεροτυπίας. Ακόμα βέβαια συζητιέται ο σχετικός, η σχετική χάρτα με εισηγήτρια την κυρία Βέμπερ και με βάση τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτιστικών όπου εισηγητής είναι ο κύριος Κόλλιν Χαιρετίζω τους δύο προσκεκλημένους μας και θα δώσω το λόγο πρώτα σε εσά κυρία Βίτα Φρέιμπερνακ και μετά στον επόμενο. Και ύστερα θα μιλήσουν οι εισηγητές και οι βουλευτές. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η έκθεση διανεμήθηκε σήμερα μόλις και στάλθηκε στα μέλη της ΕΛΕΦ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ορίστε κυρία μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών μας. Πρώτα απ' όλα το κάναμε στην Αντιπρόεδρος Επιτροπή, στην κυρία Κρού, σήμερα το πρωί. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ε, ευκαιρία που μας δίνεται να μοιραστούμε μαζί σας ε, τα βασικά σημεία αυτής της έκθεσης, γνωρίζοντας ε, το ενδιαφέρον που τρέφεται ως Επιτροπή, ε, καθώς έχετε πολλές παράλληλες δραστηριότητε στον ίδιο τομέα. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα σας εκπλήσουμε ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα αυτά, αλλά σίγουρα θα δείτε πολλά σημεία που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης, την ελευθεροτυπία και την πολυφωνία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Όταν θεωρούμε ότι η ελευθεροτυπία είναι και δικαίωση είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, πρακτικά και στην καθημερινότητα, στη ζωή σπάνια βλέπουμε την τελειότητα και βλέπουμε αποκλίσεις από το ιδανικό μιας απόλυτης ελευθεροτυπίας και μιας ποιότητας στα ΜΜΕ, όπως θα θέλαμε να δούμε. Η έκθεση μας φέρει τον τίτλο Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωση για τη διαφύλαξη της Ευρωπαϊκή Δημοκρατία γιατί εκεί εστιάζουμε. Και όπως ανέφερε και πρόεδρος, είμαστε μια μικρή ομάδα που εργάστηκε εντατικά και κατά τη διαβούλευση υφιστάμενων εκθέσεων και λοιπής βιβλιογραφίας και στις επαφές που είχαμε με άλλες ε, ομάδες ενδιαφερομένων όπως και με τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και με άμεσο διαλόγο με αυτές. Η ανησυχία μας ήταν η εξής. Θέλαμε να δούμε ποιο θα ήταν το ιδανικό. Η ιδανική κατάσταση όπου θα έχουν απόλυτη ελευθερία τα ΜΜΕ και θα υπάρχει απόλυτη πολυφωνία και όπως συμβαίνει σε κάθε πλατωνικό ιδανικό, μόνο ε, με μια προσωμείωση μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου. Δηλαδή τα έψιλον που να είναι απόλυτα ελεύθερα από οποιαδήποτε παρέμβαση ε, πολιτικών δυνάμεων ή ιδεολογιών, έψιλον που δεν υπόκειται τις ε, διαταγές των ιδιοκτητών τους και δεν έχουν γνώμονα το κέρδος των ιδιοκτητών τους, όπως και τα υλικά συμφέροντα των διαφημιστών που χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ και τα οποία εξαρτούν από τους διαφημιστές την ύπαρξή τους. Και τρίτο στοιχείο που λέμε υπόψη είναι ο ρόλος του τελικού χρήστη, του πολίτη δηλαδή, του απλού ανθρώπου που ιδίω λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για θέματα διακυβέρνησης της τοπικής κοινωνίας έως της χώρας τους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καμία επιθυμία να κάνουν προσπάθεια να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους και άρα αποστασιοποιούνται και δεν συμμετέχουν ε, στο, κοινωνικό, στο πολιτικό γίγνεσθε. Η παθητικότητα λοιπόν του πολίτη σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό ένα κίνδυνο για την δημοκρατία, αν θέλουμε να λειτουργεί καλά. Γιατί αν θέλουμε να λειτουργεί καλά η δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει ε, ενεργό συμμετοχή στα κοινά από τους πολίτες. που πολύ συχνά ούτε στις εκλογές συμμετέχουν και πολλές φορές δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στα κόμματα, αυτά που ψηφίζουν και αυτά που δεν ψηφίζουν. Εξετάσαμε λοιπόν τα προβλήματα που, έχουν, που έχουμε εντοπίσει και που θα γνωρίζετε και εσείς, τι είδους προβλήματα είναι αυτά. Και εξετάσαμε και τους τρόπους με τους οποίους οι νομοθέτες σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Ιστορικά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα παραδοσιακά μέσα, που συνήθω είναι α, τα έντυπα μέσα, τα οποία α, περνούν από αυτορύθμιση παραδοσιακά. Αν δεν υπάρχει αυτορύθμιση, θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σε μια χώρα, ότι υπάρχει λογοκρισία, προπαγάνδα, υπάρχει πλήσιμο αν θέλετε, σε αυτή τη χώρα, αν υπάρχει απόκληση από αυτή την αυτορύθμιση. Έπειτα υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα απτοκακουστικά, μέσα. Γνωρίζω ότι υπάρχει νομοθεσία και αυτά που αφορά την κατανομή συχνοτήτων και άλλα θέματα. Και πάλι εδώ θα γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και ε, διχογνωμίας. Και τέλος, αυτό που αναφέρουμε και στην έκθεσή μας είναι ότι το όλο σκηνικό των ε, ΜΕ αλλάζει με τους ρυθμούς. Ο ρόλος του διαδικτύου οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες που έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Η συμμετοχή του πολίτη, του απλού πολίτη στην επικοινωνία του με τον υπόλοιπο κόσμο. Είτε αυτό αφορά ένα στενό κύκλο φίλων, είτε αφορά μια ευρύτερη κοινότητα που συμβαίνει με πολλά ιστολόγια, blog, δείχνει αυτό το φαινόμενο ότι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην επαγγελματική δημοσιογραφία και την απλή καταγραφή απόψεων είναι πολύ δύσκολο να χαραχθούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Σε ένα παραδοσιακό επίπεδο, τα μέσα μας δίνουν το τι σημαίνει στον κόσμο, τις ειδήσει. Αυτό αφορά ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού σταθμού, εφημερίδες που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μία ψηλών τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα πρακτορία ειδήσεων ή αποστέλνουν ήδη ανταποκριτέ. Επίσης, ε, πολλές ε, φορές χρησιμοποιούν τη δική τους πινελιά μέσω του σχόλου των συνταχτών και των λοιπόν αρθρογράφων. Και ο τελικός χρήστης, ο πολίτης, ο ακροατής, ο θεατής, ο αναγνώστης έχει την τελική απόφαση. Τι να αγοράσει, ποια εφημερίδα να αγοράσει, ποιο πρόγραμμα να δει να ακούσει. Δεν μπορεί να επηρεάσει λοιπόν ο τελικό χρήστη το περιεχόμενο, αλλά μπορεί απλά να επιλέξει τι θέλει. Όμω σήμερα τα μία συλλογή είναι πιο διαδραστικά. Δηλαδή, οι δυνατότητε για τον ακροατή και τον θεατή να ανταποκριθεί άμεσα, ακαριέα, σε αυτό που βλέπεις στην οθόνη, αυτό που ακούει στο ραδιοφωνό του. Αυτή λοιπόν η δραστικότητα αλλάζει άρδιν το σκηνικό, όπως ε, και τα ε, μοντέλα επιχειρηματικότητας που επιτρέπουν ε, να επιβιώσουν τα ΜΜΕ. Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήξαμε από τις διαβουλεύσεις μας. Και αυτά είναι στοιχεία που δημιουργούν ανησυχίε στους δημοσιογραφικούς κύκλους σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, την ασφάλεια του επαγγέλματος του δημοσιογράφου. Τη δυνατότητα δηλαδή κανείς να παραμένει α, δημοσιογράφος επαγγελματίας και να βγάζεται προς το ζήν. Και να συνεχίσει αυτή την επαγγελματική πορεία, γιατί καθώς όπως στην περίπτωση των εφημερίδων βλέπουμε ότι χάνουν αναγνώστες τον ανταγωνισμό με άλλα μέσα ενημέρωσης ή υπάρχουν οι διανομής ειδήσεων μέσω του διαδικτύου που απλά ανακυκλώνουν υλικό και ειδήσει που έχει δημιουργηθεί από κάποια άλλη πηγή. Και επειδή απλά ανακυκλώνουν ειδήσει, δεν χρειάζεται να απασχολήσουν επαγγελματίε δημοσιογράφου για να το παράγουν αυτό. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα που ανακύπτουν και ένα που αναφέρουμε και αφορά τον πολίτη, έχει το εξή, ότι είναι δύο απόψει σχετικά με το τι συμβαίνει με τον πολίτη. Από τη μία ότι υπάρχει μια κάποια εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά μέσα και το διαδίκτυο, ότι δηλαδή ο πολίτης φιλτράρει μέσω του δικτύου ε, τις πληροφορίες που λαμβάνει και καταλήγει μόνο σε αυτές που επιθυμεί και μάλιστα κάποιοι εκφράσουν σαν ότι αυτό θα οδηγήσει στην απομόνωση των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στα κοινά και σε δημόσιο διάλογο. Κάτι δηλαδή που κινητοποιούσε η παραδοσιακή δημοσιογραφία. Όμως, το, δεν υπάρχει κάποιο μέσο που από μόνο του να φιλτράρει, αν θέλετε, τις πληροφορίες και τις ειδήσει. Οι δυνατότητες λοιπόν που παρέχουν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σε έναν βαθμό δίνουν στον πολίτη μια μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για το τι θέλει να καταναλώσει αν θέλετε. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν πέρα από την υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνίας στα ΜΜΕ που είναι κάτι θεωρώ δεδομένο και εσείς θα, θα πείτε κάτι παρόμοιο και η συνάδελφος θα πει κάτι παρόμοιο, το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο θα δείτε και κάποιες θέσει που καταλήγουμε στην έκθεσή μας σχετικά με το ρόλο του απλού πολίτη. Μεταξύ άλλων θέλουμε ο αλφαβητισμός των μέσων ενημέρωση να βοηθήσει γενικότερα στον αλφαβητισμό και στο να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα. Ξεκινώντας από τη μέση εκπαίδευση, καθώς είτε σε πολιτικές επιστήμες, είτε σε μαθήματα τύπου αγωγής του πολίτη, ε, οι μαθητές ήδη από τη μέση εκπαίδευση να κατανοούν αυτές τις έννοιες των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας, ελευθεροτυπίας, καθώς αυτή η γνώση θα είναι στοιχείο κλειδί αργότερα στη ζωή τους ως πληροφορημένων πολιτών. Προβάλλουμε σε μια σειρά συστάσεων. Δεν θέλω να τι απαριθμίσω. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτές όταν θα θέσετε ερωτήσεις. Θα δώσω όμως τώρα τη σκητάλη στη συνάδελφο, την κυρία Τόιπλε Μέλιν. έγκριτη ε, καθηγήτρια σε θέματα συνταγματικού δικαίου, να τη ρωτήσω, να μας πει κάποια πράγματα για θέματα της δικής της ε, αρμοδιότητας για το θέμα αυτό που πιστεύω θα ενδιαφέρουν και εσάς. Ευχαριστώ πολύ καθηγήτρια Φράιμπεργκα. Θα ήθελα να πω προς όλους τους ευρωβουλευτάς ότι η κυρία Φραϊμπέργκα δεν έχει μόνο διακεκριμένο παρελθόν ως ψυχολόγος, αλλά και ως πρώην πρόεδρος της Λετωνίας. Και εγώ δεν είμαι μόνο δικηγόρος, αλλά ήμουν και υπουργό δικαιοσύνης στη Γερμανία και πολλά χρόνια βουλευτής στο Bundestag. Οι δύο άλλοι συνάδελφοι, ο καθηγητής Μαντούρο, παραδείγματο χάρη, είναι και δικηγόρος και καθηγητής δικαίου, πολύ γνωστός, καθώς και πρώην Γενικός Εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι η ελευθερία και ο πλουραλισμός, η ελευθεροτυπία, ο ελεύθερος λόγος και ο, η έγκριτη δημοσιογραφία είναι κάτι πολύτιμο για την κοινωνία όχι μόνο των χωρών μας αλλά και ολόκληρης της Ένωσης. Γιατί ο κάθε πολίτης που ψηφίζει για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, σωστή πληροφόρηση, σε ποιοτική δημοσιογραφία και σε πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Φυσικά αυτό το δεχόμαστε, αλλά όπως είπε προηγουμένως και η Πρόεδρος, χρειάστηκε να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα που σημειώνονται στα κράτη-μέλη και είναι πολλά αυτά. Στην έκθεσή μας αναφέρονται όλα. Πρόκειται για το θέμα του τύπου και των οπτικοακουστικών μέσων των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης είναι το θίθεται το θέμα του ελευθερίας του λόγου και της ποιοτικής δημοσιογραφίας. Το θέμα δηλαδή είναι πώς θα προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι μόνο η ελευθερία του λόγου αλλά και η ελευθεροτυπία γενικότερα. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του ποιος θα είναι ο ενδιάμεσος, ποιος θα έχει τι καθήκον μεταξύ οργάνων της Ένωσης και εθνικών κρατών. Χρηματοδότηση, επιτήρηση, εποπτεία κτλ. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην έκθεσή μας. Όλα. Και καθώς εσείς είστε οι νομοθέτες, εσάς θα έπρεπε να ενδιαφέρει περισσότερο για να μπορέσετε να βασιστείτε σε αυτά τα στοιχεία και να κάνετε συστάσεις και προτάσεις, γιατί και εμείς κάνουμε 30 συστάσεις, αλλά δεν υποκαθιστούμε το έργο σας. Εσείς θα τα πάρετε αυτά, θα τα συζητήσετε, θα διαφωνήσετε, θα συμφωνήσετε και θα δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να εφαρμοστούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να σας πω και αν έχετε απορίες με τα χαράς να σας τις λύσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τις δυο σας. Τώρα, στρέφομαι στις και στους συναδέλφους. Και πρώτα η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Φράιμπεργκερ και την κυρία Υπουργό Ντόιμπλερ Γκμέλιν για την εκθεσή τους. Βρίσκω ότι είναι σημαντικό που συζητείτε τώρα το κείμενο των συμπερασμάτων τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού σύντομα θα ψηφίσουμε την έκθεση που επεξεργαζόμαστε για το standard setting για την ελευθερία του τύπου σε όλη την Ευρώπη. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω την Επίτροπο κυρία Κρούς η οποία αποφάσισε να ιδρύσει αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων για την ελευθερία του τύπου. Και ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλες και όλους για τις προσπάθειες και το έργο τους. Από πολλές πτυχές, τα πορίσματα και οι συστάσεις που μας υποβάλλεται συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό λοιπόν με το περιεχόμενο της δικής μας εκθέσεως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όντως είναι σπάνιο να βλέπει κανείς τόσο επικοδομητική προσέγγιση όπως αυτή της οποίας κατέστην μάρτης εγώ από όλες και όλους τους συναδέλφους μου που είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν την ελευθερία του τύπου. Κάποιες από τις διατυπώσεις που επιλέξατε εδώ ηχούν πολύ ευχάριστα στα αυτιά μου. Όταν λέτε για παράδειγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρηθεί αρμοδία για την προστασία της ελευθερίας του τύπου και της πολυφωνίας στο επίπεδο των κρατών μελών, αυτό για μένα είναι ακριβώς αυτό που πίστευα και εγώ όταν απεφάσισα να βλάβω την εκθέση αυτή, γιατί δεν είναι θέμα επικουρικότητας, είναι θέμα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελούν θεμέλιο όντω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά λοιπόν από τα όσα διαλαμβάνει η εκθεσή σας, ίσως βέβαια με κάπως διαφορετική φρασιολογία, θα τα βρείτε και στην έκθεση επί της οποίας σύντομα θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι εν τέλει το μήνυμα που θα συναποστείλουμε, δηλαδή και από τη δική σας ομάδα εμπειρογνωμόνων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι ένα κοινό μήνυμα που θα λέει πόσο σημαντικός ε, πόσο σημαντική υπόθεση είναι αυτή η, προστασία δηλαδή της ελευθερίας του τύπου. Θα ήθελα τώρα, αν μου επιτρέπετε, να σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις για καλύτερη κατανόηση. Ομολογώ ότι σύντομη μόνο ματιά έριξα στην εκθέσή σας, αλλά επιθυμώ να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα για την δική μου ιδίω ε, κατανόηση. Κυρίως για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ή την κρατική χρηματοδότηση. Στο, στη σύσταση σας υπαριθμούν 6 λέτε ότι το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει όπου υπάρχει αποτυχία της αγοράς και μειώνεται έτσι η πολυφωνία, η οποία πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό δημόσιο αγαθό. Τι εννοείται ακριβώς. Στην υπαρθμόν 27 σύστασή σας λέτε οποιαδήποτε δημόσια ownership των media πρέπει να για τις αυστηρούς κανόνες, να μην επιτρέπεται παρέμβαση του κράτους, ε, εσωτερική πολυφωνία και εποπτεία ανεξάρτητου οργανισμού που να εκπροσωπεί όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, όλους τους stakeholder. Μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό. Πάντως, εκτός από αυτά, το μόνο που μου μένει είναι να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας η κυρία Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στις δύο κυρίες καθηγήτριες. Εγώ ομολογώ ότι δεν διάβασα ακόμα όλη την έκθεση, αλλά έριξα μια ματιά στις συστάσεις σας. Και όπως η Ρενάτε Βέμπερ, με χαρά μου βλέπω ότι η πρώτη λέει ότι χρειάζεται περισσότερη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία των μέσων. Εσείς υποβάλλετε την έκθεσή σας στην κυρία Νέλη Κρούς, αλλά ίσως να γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως μαζί με την κυρία Ρέντινγκ, άλλη επιτροπό, αγωνίζεται εδώ και καιρό για να ξεκινήσει αυτή ας πούμε, η προσπάθεια για ε, την προστασία των ε, μέσων. Τι περιθώριο λιγμών βλέπετε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το πετύχει. Το δεύτερο που συστήνεται είναι η ουδετερότητα του διαδικτύου, ότι αυτή πρέπει να περιληφθεί στην κοινοτική νομοθεσία, να θεμελιωθεί στην κοινοτική νομοθεσία. Με non-state actors, με πολιτικούς, όλη αυτή η συζήτηση. Και την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κρούς, για την οποία συντάξατε την έκθεση, έκανε έδωσε μάλλον μια συνέντευξη στην Liberation και είπε ότι δεν θέλει net neutrality γιατί είπε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει δεν μπορεί να εξασφαλίσει μάλλον πρόσβαση στο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη με ουδετερότητα του δικτύου. Εσείς όμως λέτε να θεμελιωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ποια μπορεί να είναι η απάντηση στην κυρία Κρούς. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τις συστάσεις σας, θα προσπαθήσει να τις μεταφέρει σε νομοθετήματα, να τις, να τις περιβάλλει δηλαδή με τον ε, νομοθετικό μανδύα και από εκεί και πέρα το λόγο έχει ο κ. Σταβάρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάμβανα αυτά που είπε η κυρία Βέμπερ και η κυρία Σαρτζετίνη. Θα σας ευχαριστούμε και τις δύο για την παρουσία σας και την εξαιρετική έκθεση. Την... Διάβασα ήδη τις συστάσεις. Ε, και στο υπόλοιπο της έκθεσης ε, βρήκα πολλά ενδιαφέροντα σημεία ακαδημαϊκός, πώς θα έλεγα. Και θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, πράγματι ε, συνάδουν σχεδόν απόλυτα με την δική μας δουλειά και με την στροπολογία στην έκθεση Weber. Το μόνο που αισθάνομαι ότι λείπει στο κείμενό σας, αλλά μπορεί να οφείλεται στη δική μου γρήγορη ανάγνωση. Κάτι που ζητούμε εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο είναι η εφαρμογή του σχετικού εργαλείου για τον πλουραλισμό και την ε, πολυφωνία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο ήδη υπάρχει ως έννοια το είχε ζητήσει η Κομισιόν. Εξ όσων γνωρίζω, έχουν δαπανηθεί 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θεωρεί ότι δεν ε, μπορεί να εφαρμόσει αυτό το εργαλείο λόγω της επικουρικότητας. Η Κομισιόν, από τι απαντήσεις που μας δίνει, προσπαθεί να κάνει κάτι. Εμείς προσπαθούμε μάλλον να πιέσουμε την Κομισιόν να εφαρμόσει αυτό το εργαλείο αν έχει ήδη δαπανίσει και τόσα εκατομμύρια για τη δημιουργία του. Και η απάντηση της Κομισιόν είναι κοιτάμε στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Είναι διαγνωστικό και μόνο αυτό το εργαλείο. Εμένα δεν με καλύπτει η απάντηση. Αν θέλει κανείς να αξιολογήσει και να εκτιμήσει ε, την πολυφωνία σε ενημέρωση, χρειάζεται τέτοια ε, εργαλεία που να κάνουν μια μέτρηση. Με ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν εξάρτητο κέντρο παρατηρητήριο. Ε, θα έλεγα ότι είναι μια καλή σύσταση. Φοβούμαι όμως ότι εδώ κάτι λείπει. Υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο έχει ήδη ε, δημιουργηθεί. Έχουν δεπανηθεί κάποια χρήματα και δεν χρησιμοποιείται. Ε, κάτι μου λείπει. Θεωρώ λοιπόν ότι η υποτρένεια της ε, λογοδοσία ένα του πολίτη θα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Στο μόνο σημείο στην έκθεσή σας που θα έλεγα ότι πάει πέρα από αυτό που εγώ θα επιθυμούσα, μιλάω προ τη κατεύθυνση και θα πήγαινε και πέρα, σχετικά Ποιο είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνία, Θεωρώ ότι αυτή η ευθύνη ε, είναι κοινή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Όχι γιατί μόνο η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει η πληροφορία να είναι διεθνική, υπερεθνική αν θέλετε, αλλά πάντοτε έτσι ήταν. Το το 8ο αιώνα οι δημοκρατίες των γραμμάτων που ήταν η βάση των δικών μας δημοκρατιών ήταν ήδη οι διεθνικές. Και οι ακαδημίες κατά μεσαίωνα πάντοτε δεν περιορίζονταν από τα εθνικά σύνορα. Θεωρώ λοιπόν ότι η εξέλιξη ε, της Ευρώπης και του ε, διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο ε, πάντοτε υπήρχε και θεωρώ ότι η υπόσχεση που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ πολίτε τη Ανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση ποια ήταν. Μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε σε εμά, γιατί αυτό είναι το καταφύγιο για την ε, α, πολυφωνία, για την ελευθεροτυπία. Αν τώρα εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε Α, αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και μόνο αποτύχουν τα κράτη-μέλη, τότε μπορεί να μετατεθεί σε εμά, είναι σαν να υπαναχωρούμε σε αυτό που α, λέγαμε και να κυρώνουμε τι υποσχέσει μα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να διαβάσουμε και να ερμηνεύουμε τι τάξει συνθήκη. Λοιπόν, να σα φαίνεται τώρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια αυτή που επέλεξα. Στι τάσει εσεί λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα αρμόδια, να αναλάβει δράση και να προστατεύσει την ελευθεροτυπία και την πολυφωνία σε επίπεδο κράτου μέλου. Ναι. Ε, είναι κάτι που το έχουμε πει και ξαναπεί και εμεί πολλέ φορέ. Σας ευχαριστώ επίσης γιατί και εσείς επιβεβαιώνετε ότι είναι πολύ σημαντικό και ισχυρό αυτό το επιχείρημα. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ είναι ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα ε, και των κρατών μελών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσουμε την ελευθεροτυπία. Κατά τα λοιπά κάνετε μια πολύ καλή δουλειά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σίπελ. Όσοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό, καλά θα είναι να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση των δύο καθηγητριών σαν βάση για μια ευρεία συζήτηση. Η ιδιαίτερη αξία της εκθέσεως συνίσταται στο ότι αυτή καθιστά σαφές ότι η ελευθερία των μέσων και επομένως η πολυφωνία και εν μέρη και η λειτουργία της δημοκρατίας μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο από πολλά και διάφορα πράγματα, όχι μόνο κρατική παρέμβαση, αλλά και οικονομικές δυσχέρειες, ιδίως μάλιστα με τα νέα μέσα, αυτά δίνουν και ιδιαίτερο ρόλο στους πολίτες. Με την εμφάνιση των λεγόμενων νέων μέσων, προκλήθηκε και μια εφορία, σαν επιτέλους τώρα όλοι οι πολίτες να είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίε. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι αυτόματο, δεν χρησιμοποιούν όλες και όλοι τις, ε, την ελευθερία αυτή πρόσβασης για να πληροφορούνται, για να ενημερώνονται για κοινωνικά θέματα ας πούμε κτλ. Αλλά πολύ συχνά και για παιχνίδια ή για ψώνια κτλ. Ω ευρωπαϊκός δρόμος, και αυτό είναι σημαντικό για μένα, γιατί το περιλαμβάνεται και σε μία από τις συστάσεις σας, είναι η αρμοδιότητα για τα μέσα. Η ερώτησή μου είναι, ποιες δυνατότητες θεωρείτε ότι έχουμε εμείς ως ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι θυμούμε τους τελευταίους μήνες να έχουμε συζητήσει συχνά το θέμα αρμοδιότητα για τα μέσα σε συνδυασμό με διάφορες οδηγίες και σε κάθε περίπτωση χρειάστηκε να περιοριστούμε στο να συστήσουμε στις χώρες μέλη να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα. Όχι μόνο δηλαδή τον τεχνικό χειρισμό των μέσων, αλλά και ποιος προσφέρει πληροφορίες μέσω των μέσων πόσο αξιόπιστος και αξιόπιστες είναι αυτές και ούτε καθεξής. Ζητούσαμε λοιπόν από τις χώρες μέλη να ενδιαφερθούν, διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Και με ενδιαφέρει λοιπόν, εάν σκεφτήκατε κι εσείς να πείτε ότι εφόσον δεν υπάρχει αρμοδιότητα αυτή, τότε πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν το διάβασα και ολόκληρο το κείμενό σας, αλλά είναι άρα γι' αυτό κάτι το οποίο προκύπτει από τις συζητήσεις με τους διαφόρους φορείς. Ευχαριστώ, Νταρόκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Νομίζω δεν υπάρχει δεν, νομίζω δεν υπάρχει ε, λετωνική καμπίνα. Καλά, παρόλα αυτά επιτρέψτε μου μια, πω μια φράση. στα λετωνικά, αλλά απευθύνεται στην κυρία Φρέιμπεργα που μιλεί την ίδια γλώσσα. Τι είπα, τι είπα, μόνο, συνεχίζει η κυρία Σδάνοκα, ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω την πρώην πρόεδρό μας εδώ παρούσα στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών. Θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για τις συστάσεις αυτές. Ακόμα δεν πρόλαβα να τις διαβάσω όλες. Όμως παρόλα αυτά έχω μερικές ερωτήσεις. Ιδίω για ένα θέμα που το βλέπω στη σελίδα 7 για την ανεξαρτησία των ρυθμιστών ή των ε, media councils. Νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είπατε και εσείς ότι είναι πρόβλημα. Το είδαμε άλλωστε σε ορισμένες χώρες μέλη και πρόσφατα. Έχετε άραγε πιο συγκεκριμένε συστάσει, πώς να εξασφαλιστεί η πολυφωνία αυτή και η ανεξαρτησία και η εκπροσώπηση όλων των, όλου του φάσματος της κοινωνίας μέσα σε αυτά τα συμβούλια, συμβούλια τύπου, που γνωρίζουμε ότι τα πιο συχνά διορίζονται από τα κοινοβούλια, χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης όλων των διαστρωματώσεων της κοινωνίας. Εγώ σκέφτηκα ίσως και απευθείας εκλογή των συμβουλίων αυτών. Με γενικές εκλογές ενδεχομένως, όπως οι βουλές. Τι νομίζετε. Ευχαριστώ κυρία Ιώτοβα. Θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και εισηγητρίες Αναμένουμε τη μελέτη αυτή από καιρό για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε και απόψεις για τα διάφορα προβλήματα που περιλαμβάνεται εκεί. Είμαι βεβαία ότι δουλέψατε σκληρά για να συντάξετε αυτές τις 40 σελίδες συστάσεων. Μετά από τις αναλύσεις σας, εν τέλει ποια είναι τα συμπεράσματά σας. Μπορούμε να καθιδρύσουμε πανευρωπαϊκούς μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την διαφάνεια των μέσων. Ερώτημα που συχνά θέτουν οι δημοσιογράφοι καθώς και προσωποι μη κρατικών οργανισμών. Και δεύτερο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς που να ελέγχουν την συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, γιατί η συγκέντρωση είναι απολυταρχικό φαινόμενο, είναι δικτάτη μέσα στα πλαίσια των μέσων. Κύριε Παπα-Νικολάου, επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω τις διακεκριμένες ομιλήτριες. Το θέμα σας είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα περισσότερο εάν συνδέσουμε τα όσα μας είπατε με τις βιογραφίες σας. Εγώ ακούγοντά σα, σκέφτηκα ότι οι συζητήσει που κάνουμε σήμερα εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο εθνικό για την leadership που χρειαζόμαστε και πώς αυτή η ηγεσία δράει αντιδρά σήμερα, πώς από την άλλη μεριά συμπεριφέρονταν οι ηγέτες στι δεκαετίε του 60 και του 70 και σε ποια περιβάλλοντα, διότι τώρα πιστεύω ότι και τώρα έχουμε ηγέτες, αλλά δρούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα με όλα αυτά τα media, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν και όντως σήμερα αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις αλλά και στο παρελθόν είχαμε προκλήσεις και πιστεύω ότι πριν από μερικές δεκαετίες οι τότε συνάδελφοί μας συνομιλούσαν όπως εμείς για τις προοπτικές, για τα επόμενα βήματα που θα εξασφάλιζαν την πολυφωνία, την ποιότητα των δημοκρατιών, την ελευθερία του λόγου. Και όταν έχουμε μπροστά μας όλη αυτή την ευρεία εικόνα, συμφωνώ απόλυτα με την υπαρθμότητα και νέα σύστασή σας που λέτε ότι η αλφαβήτα των μέσων πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία να έχουμε Ευρωπαίους πολίτες που να γνωρίζουν, να μπορούν να αντιλαμβάνονται την ποιότητα της ενημέρωσης, είτε αυτή προέρχεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους ή άλλους που την διοχετεύουν, όπως είπατε. Η γενική ερώτηση, η ερώτηση μου μάλλον είναι πολύ γενική. Πιστεύετε ότι οι προοπτικές μας βελτιώνονται ή ίσως όχι. Είστε αισιόδοξε. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου και τώρα επανέρχομαι στις δύο προσκεκλημένες και πρώτα την κυρία Φρέιμπεργκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη ευθύς εξ αρχής αν δεν απαντήσω στο κάθε επιμέρους σημείο ε, και αν το επιθυμείτε μπορείτε να μου το επιθυμήσετε. Πιστεύω ότι ουσιαστικά συμφωνούμε Ω προσωπός νοούμε τι αρμοδιότητε που υπάρχουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασίζονται στις ίδιες θεμελιώδεις ε, αξίες και που είναι αυτές που μας έφεραν κοντά ούτως ή άλλως και δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, αποσύνδεση αυτών. θεωρώ ότι αυτό είναι και το πλέον βασικό και κέριο μήνυμα που προσπαθεί να περάσει η εκθεσή μας. Ο ρόλος που παίζουν τα ΜΜΕ σε μια καλά λειτουργούσα δημοκρατία είναι το θέμα μας. Μετά, οι αρμοδιότητες του καθενός είναι ένα θερμό ζήτημα. Ο καθένας μας, στο καθένα μας αναλογεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι θεμελιώδες ε, αξίες ε, τη χάνουν σεβασμού. Άρα υπάρχει και αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο και επισημαίνουμε στην εκθεσή μας ότι υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι της επικουρικότητας ε, ε, δείχνει προς τα κράτη-μέλη. Ξέρετε, δεν είναι μια ομοιογενής, ομοιόμορφη κοινότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μεγάλη ποικιλομορφία, ε, μεγάλες διαφορές, πολλές γλώσσες καλύπτει, πολλές διαφορές ε, που οφείλονται στην ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη των λαών της. Και αυτό που προσπαθεί να καλύψει η αρχή της είναι η διασφάλιση αυτής της ποικιλομορφία. Και να τηρήσουμε από την άλλη να σεβόμαστε κάποιες θεμελιώδεις και κοινέ αξίες. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σίγουρα μπορείτε να πείτε τρόπο την είστε θεματοφύλακε από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, θεματοφύλακες λοιπόν των θεμελιωδών αυτών αξιών. Και δεν θα πρέπει κατά τύχη, αν θέλετε, να καταλήξουμε σε κάποια αποσύνδεση και απόκληση από αυτά τα ιδανικά. Σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζουμε ότι πάντοτε κάποιος θα τη δράσει, ένας πολίτης, μια μη κυβερνητική οργάνωση, αν όχι μια κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Κάποιος πάντοτε θα ε, στήσει το παράστημά του από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα, πιο συγκεκριμένα, κυρία Βέμπερ, μίλησε για τις συστάσεις. Σύσταση 26. 26 και 27 συγκεκριμένα. Κάπου τις είχα. We have tried. We have tried to... Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές που μας διέπουν χωρίς να μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. ευχαριστώ πολύ, Χέτα, που μου δίνει το κείμενο. Σε γενικέ γραμμές προσπαθούμε εδώ να ορίσουμε τις γενικές αρχές. Πρώτα απ' όλα, η γενική αρχή τη σύσταση 26 είναι η εξή. Πέρα από το κέρδος, ποιες άλλες αξίες υπάρχουν στην κοινωνία και πώς θα τις ασφαλίσουμε. Διότι αν πάντοτε ο γνώμονας μας είναι το κέρδος και αν το επιχειρηματικό πάντοτε μοντέλο υπερέχει, και μόνο τα ΜΜΕ που δίνουν κέρδος στους ιδιοκτήτες τους ε, επιβιώνουν, τότε θα πρέπει ο μισός κόσμο να μιλά αγγλικά και μας ως κινέζικα και να τελειώνουμε. Θα χάσουμε όλες τις υπόλοιπε γλώσσες και τους ε, πολιτισμούς μας, ε, τις επιμέρους ε, διαφορές μας και πόσα άλλα στοιχεία πολιτισμού που θα εξαφανιστούν. Μιλάμε για πολιτισμικές ε, αξίες στην κοινωνία που δεν ε, αποδίδουν υλικά ωφέλη αναγκαστικά. Είναι όμως αξίες ε, σημαντικές για κάποιες πτυχές κοινωνίας, για κάποιους τομείς κτλ. Για παράδειγμα, λέγαμε, ποιο είναι το ποσοστό των ακροατών ραδιοφώνου που ακούει κλασική μουσική. Ε, εκπλήσει και πόσο χαμηλό είναι αυτό το ποσοστό. Αν λοιπόν το κίνητο ήταν καθαρά οικονομικό θα πρέπει να εξαφανιστεί από τις αδειοσυχνότητε η κλασική μουσική και θα ήταν μια τεράστια απώλεια πιστεύω. Κάτι τέτοιο είχαμε υπόψη. Επιτών μιλάμε για αυτορύθμιση ε, των ΜΜΕ ε, και οι ενώσεις των μέσων ενημέρωσης. Αυτές οι ενώσεις είναι ένας ενδιάμεσο ανάμεσα στην κοινωνία ε, πολιτικής, από την άλλη πολιτικών μάλλον, των πολιτικών και των ιδιοκτητών τους, γιατί και οι ιδιοκτήτες θέλουν μέσω της ιδιοκτησίας τους, τα ΜΜΕ, κάτι να κερδίσουν, να κερδίσουν προς το Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των τριών. Και μια άλλη σύσταση που αφορά το ζήτημα αφορά αυτές τις ενώσεις ε, ε να είναι όσο γίνεται ανεξάρτητα. Και όπως ρωτήσατε, αυτό οφείλ, μάλλον ξεκινά από τη σύνθεσή τους. Η, επιλογή των μελών πολλές φορές ε, γίνεται μέσω των κοινοβουλίων και τα κοινοβούλια μπορούν να διασφαλίσουν τη δημοκρατία και άρα την συμμετοχή και την εκπροσώπηση όλων, αν θέλετε, των φωνών α, της κοινωνίας. Τεχνικά όμως, τεχνικοί κανόνες που να διασφαλίζουν αυτή την ισορροπία. Για παράδειγμα, να λες κανόνες που να λέει ότι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να εκλεγεί αυτή η ένωση μέσω του τύπου. Και ότι η ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να διασφαλίσει επαρκή ποικιλία απόψεων σε αυτή την ένωση τύπου. Όμως πολύ συχνά μπορεί να συμβεί σε διάφορες χώρες. Ε, τελικά είναι πολύ μονοφωνική και μονομερή η εκπροσώπηση σε αυτές τις ενώσεις. Το θέμα είναι να βλέπουμε ποιος είναι ο απότερος σκοπός των ρυθμίσεων που επιβάλλουμε και ποιο, τι καλύτερα να εξυπηρετήσει ένα οποιοδήποτε όργανο ε, ζητούμε να συσταθεί. Και άρα θα πρέπει να δημιουργούν του κατάλληλους κανόνες, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό το σκοπό. ώστε να μην νομοθετούμε απλά, να μπορούμε να επιτύχουμε και τους σκοπούς μας στην πράξη. Τώρα, η συγκέντρωση μέσω ενημέρωσης ε, και η σχετική νομοθεσία, κάτι πολύ ε, ενδιαφέρον. θίξαμε σε αυτό το θέμα, θα έλεγα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα από μόνο του. Γνωρίζετε κι εσείς ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Προσωπικά έχω την αίσθηση ότι αν σε μια χώρα, αν κάθε εφημερίδα είναι στα, αρχαία, στα, είναι στα χέρια ε, του ίδιου μήλου, ε, ε, αυτό δεν είναι η κατάσταση ούτε για την πολυφωνία, ούτε για την ελευθεροτυπία. Ακόμα, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία από επιρροές ε, της δημοσιογραφίας. Α, η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας είναι ένα ζήτημα. Οι κώδικες δεντολογίας που πρέπει να ακολουθούν, ναι. Η διαφάνεια θα πρέπει δηλαδή αυτέ οι βασικέ αρχέ, της εντοντολογίας και διαφάνεια να υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Αλλά από εκεί και πέρα, κομμάτι τη δημοκρατία είναι και οι πολιτικές θέσεις, Πολιτικέ απόψει. Αρκεί κανεί να εκφράζει τι πολιτικέ του απόψει, ώστε να μπορεί κανεί να διακρίνει ε, τι είναι ένα γεγονό, μια είδηση και τι είναι μια άποψη, μια γνώμη. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Εγώ είμαι στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι το μέλλον μπορεί να πάει το καλύτερο γιατί έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε, να επηρεάσουμε τα πράγματα ώστε το μέλλον να καλύτερο. Οπότε καλό και εσά, ε, ε, τους κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτές. Από εσά εξαρτάται. Από την δική σας ενεργητικότητα και ικανότητα να κάνετε κάτι για να επηρεάσετε το μέλλον και βεβαίω να αποτανθείτε και στου πολίτε που πρέπει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, όπω είπα και νωρίτερα, πράγματι μπορεί η ηλεκτρονική δημοσιογραφία μπορεί να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να διευρύνει τι γνώσει του, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει το ίδιο εργαλείο για να απομονωθεί και να συρρυκνώσει τελείω τι γνώσει του. Δηλαδή, μπορεί κανεί να βλέπει το διαδίκτυο για να παίζει παιχνίδια ε, και μόνο. Ε, εξαρτάται λοιπόν από, το, από τον κάθε χρήστη και από τον κάθε πολίτη το πώς χρησιμοποιεί ένα τέτοιο εργαλείο. Ελπίζω να απάντησα στα βασικά ερωτήματα και η συνάδελφο θέλει να συμπληρώσει. Only for one minute, because then I have to... Ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι μόνο, γιατί πρέπει να πάω αεροπλάνο. Ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε τις συστάσεις που κάναμε λεπτομερέστερα, γιατί θα δείτε ότι Μερικές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Σας κατευχαριστώ κυρία Βέμπερ που είπατε ότι συμφωνούμε βασικά. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό. Βέβαια και εμείς διαβάζουμε πάρα πολλές εκθέσεις δικές σας και του Συμβουλίου της Ευρώπης από οργανώσεις και από δημοσιογράφους τα βλέπουμε όλα και τα βάλαμε όλα στην έκθεσή μας. Ήθελα μόνο να τονίσω ότι τις συστάσεις αυτές δεν τις κάνουμε μόνο για να χαρείτε, αλλά θέλουμε και να σας προκαλέσουμε να αντιδράσετε νομοθετικά, γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερες δικαιοδοσίες, αλλά δεν το λέμε στις συστάσεις αυτό ούτε προς την Επιτροπή, προς την Κομισιόν. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που πρέπει να το πούν. Αλλά είναι απαραίτητο να αποσαφινιστεί ότι το άρθρο 11 της χάρτας, λέει ο ομιλήτρια, είναι σαφές. Το θέμα δεν είναι ότι με την επικουρικότητα θα γίνουν όλα. Το θέμα είναι πώς. Αν έχετε το χρόνο λοιπόν κοιτάξτε τις συστάσεις μας, είναι ευνόητες και εύληπτες. Και τότε να ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Φράιμπεργα και κυρία Γκμέλιν για την προσέλευσή σας και για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Τώρα το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα. Προστασία δεδομένων. Στην περασμένη συνεδρίαση της ΕΛΕΦ στις 10 Ιανουαρίου οι εισηγητές Δρούτσας και Άλμπρεχτ υπέβαλαν το πρώτο σχέδιο έκθεσής τους. Έγινε μία ανταλλαγή απόψεων και λόγω του ενδιαφέροντος των μελών της Επιτροπής συμφωνήσαμε να γίνει και δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης σήμερα, που αν δεν απατώμε είναι 21 Ιανουαρίου. Προτείνω λοιπόν και τα δύο σχέδια έκθεσης, τα δύο σχέδια έκθεσης να τα εξετάσουμε χωριστά για να δούμε τι ακριβώς έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Πρώτα λοιπόν η έκθεση του κύριου Δρούτσα για την οδηγία για την προστασία των δεδομένων και πρέπει να φύγει πριν λήξει η συνεδρίαση και μετά θα δούμε την έκθεση του κυρίου Αλμπρίχτ παρακαλώ τους συναδέλφους να σχολιάσουν το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Δρούτσα και την οδηγία που εξετάζει βέβαια. Η, κατάθε, η διορία για την κατάσταση των απολογιών λήγει στις 27 Φεβρουαρίου. Στην περασμένη συνεδρίαση έγινε λόγος για παράταση η πλειοψηφία συμφώνησε να τηρηθεί η ίδια διορία που είναι ήδη πολύ, είναι δύο μήνες. Και αν το Κοινοβούλιο θέλει να καταλήξει σε συμφωνία μέσα στο 2013 πρέπει να αρχίσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Προς στιγμή λοιπόν διατηρείται η διορία ως 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Α, υπάρχει και μία πρόσθετη ανακοίνωση. Προσθετή. Μας ζήτησαν να επιτρέψουμε την είσοδο κινηματογραφιστών εδώ για να κινηματογραφήσουν τη συζήτηση. Έχουν έρθει και άλλες φορές. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, να έρθουν. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή κύριος Δρούτσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα στην προηγούμενη μου παρουσίαση, απλώς έτσι διαδικαστικά να σας προτείνω τα εξής. Είπατε από την αρχή ότι πρέπει να δούμε την κάθε τις δύο εκθέσεις χωριστά. Σωστό, πολύ σωστό. Αλλά για δύο λόγους ίσως πρακτικότερο θα ήταν να ξανασυζητηθούν μαζί. Πρώτον, γιατί για μας είναι σημαντικό να θεωρηθεί δέσμοι, να θεωρηθούν δέσμοι και τα δύο και δεύτερον διότι οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για το γενικότερο πρόβλημα άρα του κανονισμού και τρίτον και να σας πω to Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά βλέποντας εδώ στην αίθουσα δεν διαπιστώνω την παρουσία και πολλών συναδέλφων που να μπορούν να μιλήσουν και εμείς τη αιτήση των υπολείπων προβλέψαμε αυτή τη δεύτερη συζήτηση για το σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως ελπίζω να έρθουν κι άλλοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πάντως έχοντας συνεννοηθεί και με τον Γιάννα Άλμπρεχτ ξαναπροτείνω μήπως οι συνάδελφοι όταν θα μιλήσουν να αναφερθούν και στις δύο εκθέσεις, αν θέλουν, αν θέλουν. Στο κυρία Ζήπερ. Ευχαριστώ. Θα ε, μιλήσω εγώ για την οδηγία, γιατί ο Γιάννα Άλμπρεχτ δεν μίλησε ακόμα επισημαίνω και εγώ τα όσα εξήγησε ο κύριος Δρούτσας στην τελευταία συνεδρίαση, διεξήχθη αρκετά έντονη συζήτηση για το ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για συζήτηση και καλά θα ήταν παρόλες τις ενδεχόμενες δυσχέρειες που μπορεί να έχει ο καθένας να είναι περισσότερες και περισσότεροι συνάδελφοι εδώ παρόντες και παρούσε σήμερα για να γίνει πιο εκτεταμένη συζήτηση. Βέβαια είναι σωστό και εξακολουθώ να το υποστηρίζω ότι και τα δύο αυτά έγγραφα, δηλαδή και την οδηγία και τον κανονισμό, πρέπει να τα εξετάσουμε μαζί, όσο είναι αυτό δυνατό, ως δέσμοι. Και μάλιστα και επί του ουσιώδους περιεχομένου υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις μεταξύ των κειμένων. Παρ' όλα αυτά, μου φαίνεται σωστό να ξανασυζητήσουμε διεξοδικά για την οδηγία. Διότι στην εντύπωση της κοινή γνώμης, ο κανονισμός είναι αυτός που κατησχύει και η οδηγία κάπως υστερεί. Βεβαίω έχει μεγάλη σημασία ο κανονισμό, αλλά θεωρώ ότι και η οδηγία είναι το ίδιο σημαντική για όσους κάποτε θα φυγούν από το θέμα και θα θέσουν το ερώτημα πόσο προστατευμένα είναι τα δεδομένα μου όταν δηλαδή θα έχουν θέματα δικαιοσύνης κλπ. Και ο φόβος μου προκειμένου είναι ότι για να συζητήσουμε από κοινού και τα δύο ίσως τελικά να θυσιαστεί κάπως η οδηγία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω και τους δύο εισηγητές να μην τάσσονται μόνο υπέρ του χαρακτήρα πακέτου δέσμης, αλλά να τονίσουν και τα ιδιαίτερα στοιχεία των δύο εγγραφών. Επειδή λοιπόν είναι πολύ λίγοι οι παρόντες και παρούσες, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα και ιδίω όσον αφορά την οδηγία. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί και πάλι ποια είναι τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας. Και να τονιστεί και πάλι ότι γενικά τα δεδομένα αυτά σε ποινικέ διαδικασίες ή από ανακρίσεις κλπ. πρέπει να προστατεύονται. Διότι αφενός διαδικασία που αρχίζει στο εθνικό επίπεδο αργότερα λαμβάνει διασυνοριακό χαρακτήρα. Και τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να αποθηκεύονται δεδομένα και μετά από, το, από την περάτωση της διαδικασίας και ενδεχομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ή να διοχετευθούν διασυνοριακά, διαμεθοριακά σε άλλες αρχές. Εκεί χρειάζεται λοιπόν να συνταχθούν κάποιες προδιαγραφές. Εγώ είπα ότι αυτό δεν πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ανακρίσεις, στις ποινικέ ανακρίσεις, γιατί και οι διεξαγόντες της έρευνας έχουν ενδιαφέρον να τηρείται η προστασία των δεδομένων. Αλλά και το δικό μου προσωπικό ε, ενδιαφέρον με ποιον τρόπο δηλαδή θίγομαι από μια ποινική διαδικασία, αυτή την ερώτηση τη θέτει και ο κάθε πολίτης, είτε ως κατηγορούμενος είτε ως μάρτυρας σε μια ποινική διαδικασία. Έχει λοιπόν κάθε ενδιαφέρον και συμφέρον να μην έχει ο καθένας πρόσβαση σε κάποια δεδομένα. Να τη χάνουν λοιπόν αυτά υψηλής προστασίας. Πρέπει λοιπόν να ξαναθέσουμε το ερώτημα της χρήσης των αποδεικτικών στοιχείων και της προστασίας τους. Και θα χαρώ βεβαίως εάν σε κάποια μελλοντική ευκαιρία ή το αργότερο όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες να συζητήσουμε και τις πτυχές αυτές. Το ίδιο όπως και τα άλλα ουσιαστικά και σημαντικά στοιχεία της, ε, του κανονισμού. Ευχαριστώ κύριος Βόση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και τόσο διαφορετικές από αυτές που είχα ακούσει την προηγούμενη φορά. Θα αρχίσω με την οδηγία. Στον τομέα της οδηγίας, αυτό που επιδιώκουμε είναι η ασφάλεια δικαίου. Καθώς και η εμπιστοσύνη στην χρήση των στοιχείων και όλων των εμπλεκομένων αρχών, ποινικών αρχών. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς θεωρούμε ότι το θεμελιώδε δικαίωμα προστασίας των δεδομένων και της προσωπικής σφαίρας πρέπει να προστατεύεται από το ίδιο το κράτος απέναντι σε οποιαδήποτε κατάχρηση των δεδομένων αυτών. Ειδικά τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες ποινικών υποθέσεων αλλά και την εκτέλεση ποινών, η προστασία δεδομένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλες σημαντικές ιδέες της βασικής θεωρίας που προκύπτει από το κρατικό μονοπόλιο της εξουσίας. Για παράδειγμα, την ε, διασφάλιση της γενικής ασφάλειας, τις έρευνες σε ποινικέ υποθέσεις και ούτω καθεξής, τα οποία πρέπει να εναπόκεινται στο κράτος. Και βεβαίως πρέπει το κράτος να εξασφαλίζει ότι τα καθήκοντα αυτά τα εκτελεί το κράτος και προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Εγώ δεν κουράζομαι να λέω ότι ειδικά για την αστυνομική και, δι... δικανική συνεργασία υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ενόμων τάξεων των γειτονικών άλλωστε χωρών μελών της Ένωσης. Ώστε εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερα ευαίσθητη προσέγγιση και μέσω ευρωπαϊκών ρυθμίσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαφορές, αλλά οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν με μεγάλη ευαισθησία και πολύ σταδιακά. Γι' αυτό για το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 16 της συνθήκης δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το ενδεχόμενο αντιφασκουσών δικαστικών αποφάσεων. Και εκεί χρειάζεται να ισχύσει ρεαλισμός. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάγκη εξισορρόπησης της ανταλλαγής πληροφοριών. Και στο 16 παράγραφος 2 πάλι της συνθήκης εργασίας της, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρμοδιο... Ε, αυτά εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Όμως, μπορεί να υπάρχει και συνεργασία, αστυνομική συνεργασία που δεν μπορεί όμως να βασίζεται μόνο στο άρθρο 87 της συνθήκης, γιατί υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα της προστασίας των δεδομένων που λειτουργεί οριζόντια και μπορεί επομένως να επισέρχεται και σε τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν σε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ενδεχομένως να παραβιάζουν την αρχή της ευικουρικότητας. Γι' αυτό και στα πλαίσια βέβαια της, θέσης, της ε, γραμμής της πολιτικής μου ομάδος, εγώ πιστεύω ότι μέσα σε αυτή την οδηγία πρέπει να καθιδρυθούν ελάχιστες προδιαγραφές. και νομίζω ότι η διαμεθοριακή αυτή ανταλλαγή δεδομένων εν τέλει θα πρέπει να υπόκειται σε ελάχιστες προδιαγραφές, σε ελάχιστα στάνταρτ για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία. Πρέπει αφενός να ενισχυθούν τα δικαιώματα του ατόμου και καλά το καταφέραμε νομίζω και πολύ καλά τα κατάφερε ο εισηγητής και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε τις αρχές της διαφάνειας και του ελέγχου και πώς αυτές οι αρχές θα θεμελιωθούν στον τομέα αυτό. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια και τον στόχο της προστασίας και της προστασίας της ασφάλειας δηλαδή και της δίωξης των ενδεχόμενων εγκλημάτων. Το δικαίωμα δηλαδή της προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Εγώ πιστεύω ότι ήδη μέσα στην οδηγία πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Στο κεφάλαιο 1 λέγουμε ότι πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογή και η άποση του κινδύνου, η αντιμετώπιση του κινδύνου. Και γι' αυτό οι χώρες μέλη πρέπει να υπερβούν εν προκειμένου τις ελάχιστες προδιαγραφές, έτσι ώστε η οδηγία να μην είναι να μην ε, ακολουθεί το στόχο της εναρμόνισης παρά μόνο των ελάχιστων προδιαγραφών όπως είπα και πριν. Και όπως έχουμε ξανασυζητήσει, το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί στα όργανα και άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κεφάλαιο 2, νομίζω πρέπει εδώ οι μεγάλοι τομείς όπως ε, προστασία των δεδομένων κλπ. πρέπει να προσαρμοστούν στο κείμενο της συνθήκη. Το άρθρο 5 πρέπει να δούμε την γραφειοκρατία και το προκαλούμενο κόστος. Ο στόχος της προστασίας δεδομένων εδώ είναι δεσμευτική αρχή της ποινική προστασίας και γι' αυτό νομίζω ότι τα άρθρα 6 και 7 πρέπει να τα επανεπεξεργαστούμε σε ό,τι αφορά δηλαδή τον δεσμευτικό σκοπό και για την χρήση δεδομένων από άλλες χώρες μέλη. Εδώ πρέπει να διευρυνθεί το άρθρο 13. Στο κεφάλαιο 3, σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα της ατομικής του, του θυγωμένου ατόμου δηλαδή, εδώ έχουμε ανάγκη περιορισμού στο άρθρο 12 με εξισορρόπηση της ε, ανάγκης προστασίας με την ανάγκη παροχής πληροφοριών. Το δικαίωμα για πληροφορίες στην καταγραφή των δεδομένων όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Νομίζω αυτό περιτέμνεται και σε ό,τι αφορά τέλο το δικαίωμα τη διαγραφή ή τη διορθώσεω των προσωπικών δεδομένων και το κείμενο αυτό πρέπει να επανεξεταστεί και να διορθωθεί. Στο κεφάλαιο 4 θα προσπαθήσω να είμαι ε, συντομότερο γιατί θέλω να μιλήσω και για τον κανονισμό μετά. Στο άρθρο 23 με τα έγγραφα και επίσης και έχουμε και το άρθρο 10 της αποφάσεως πλαίσιο του 2008 και πρέπει αυτά να συνεξεταστούν και ίσως να γίνει το κείμενο εδώ κάπως πιο αυστηρό. Στο άρθρο 27 πρέπει να παραπέμψουμε στο άρθρο 22 της ε, αποφάσεως πλαισίου και να κάνουμε και τη σχετική προσαρμογή και με τις ε, κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις έχουμε μιλήσει ήδη και στα πλαίσια του κανονισμού προστασίας των δεδομένων. Πρέπει να περιοριστεί λίγο αυτή η μετακίνηση αρμοδιοτήτων. Αυτά είναι λίγα από τα σχόλια που έχω να κάνω. Έχω και άλλα, αλλά ενδεχομένως ε, σε άλλη χρονική στιγμή. Αυτά για την οδηγία. Κύριε Σαντσίου, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι ε, θα έλεγα ότι κάλυψαν τα πιο πολλά από τα θέματα που ήθελα και εγώ να αναφέρω και για τις δύο εκθέσεις. Οπότε θα επιμείνω σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Το γεγονό τεχνολογική πρόοδο ε, μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε όλο και πιο πολλά δεδομένα. Αυτό σημαίνει την αναγκαία και αυτή η αποθήκευση. Η αποθήκευση θα πρέπει να περιορίζεται με βάση συγκεκριμένου κανόνες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ευρεία συνειδητοποίηση μεταξύ των πολιτών ότι αποθηκεύονται τα δεδομένα τους, άρα και θα πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί οι πολίτες, επίτευνα να έχουν πιο υψηλό επίπεδο υπευθυνότητα με ένα θεσμικό πλαίσιο προσεδεδομένων ε, που θα αναλάβουν ε, οι αρχές προστασίας δεδομένων, ώστε να έχουμε την ορθή εφαρμογή των δύο νομοθετικών εργαλείων, κανονισμού και οδηγίες. Θα πρέπει να οριστεί επίσης η νομοθετική πράξη ότι η αποθήκευση και η χρήση αυτών των δεδομένων δεν θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, αλλά μόνο όταν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη ανάγκη και απόδειξη αυτής. Και όταν αποδεικνύεται η ανάγκη αυτή, το, ο όγκος των αποθηκευόμενων δεδομένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το απόλυτα αναγκαίο. Και εδώ μιλάμε για την χρήση αρχών, δημόσιων αρχών όπως και ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων κτλ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη χρήση του καθενός. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούν ούτε, και το χειρότερο είναι να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς ε, προτέρα έκριση. Οι πολίτες επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει αποθήκευση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων, να υπάρξει εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών ακριβώς γύρω από αυτό το ζήτημα και καθόλου αυτή την αλυσίδα αποθήκευση, χρήση και μεταβίβαση δεδομένων, να υπάρχει σαφή γνώση και κατανόηση από πλευρά των διαφερόμενων τι σημαίνει αυτό για τα δεδομένα του κατά τη συλλογή και μετά ε, των δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε έλεγχος ως προς το πώς χρησιμοποιούν οι αρχές που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούν αυτά. Από εκεί πέρα, στι ε, δύο εκθέσει, βλέπω μια πρόοδο προσωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ανέφερε, όμω, πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο αυτά τα σημεία και με τι τροπολογίε που έχω υποβάλει ελπίζω να υπάρξει βελτίωση αυτών. Ο σύντομη παρατήρηση πρώτα. Σίγουρα όλα αυτά τα χιόνια έχουν εμποδίσει κάποιους να προσέλθουν και εγώ καθυστέρησα. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να συζητήσουμε. Και εγώ θα τοποθετηθώ πρώτα για την οδηγία. Βεβαίω θα συζητούμε αυτά σε ένα θέμα τη ημερήσια διάταξη και τα δύο αυτά κείμενα. Για την οδηγία έχω την εντύπωση ότι ω Ευρωκοινοβούλιο δεν καταλήξαμε στον τελικό μας στόχο, δηλαδή μια καταρχήν ενιαία αρρύθμιση της προστασία του δεδομένου. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι στον πρώην τρίτο πυλώνα, δηλαδή αστυνομική και δικανική συνεργασία, οι προσεγγίσεις είναι πολύ διαφορετικές. Η προτινόμενη οδηγία εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτέ τις διαφορές αυτές στον τομέα αστυνομίας και δικαιοσύνης. Και εξαιρούνται πάλι εδώ οι ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές κλπ. Κάτι το οποίο ήδη επικρίναμε. Και από την άλλη μεριά, μυστικές υπηρεσίες και διάφορες υπηρεσίες κρατικής ασφαλείας, διότι εκπίπτουν τις αρμοδιότητες αυτής. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κοινούς κανόνες. Αν σκεφτούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στα πλαίσια της ε, σύμβασης του ΠΡΙΜ ή της συνεργασίας των αρχών στον τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπόλ για την ανταλλαγή δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε κανόνες κοινού. Αφετέρου μιλούμε εδώ για βασικές αρχές θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν σκεφτούμε πώς εργαζόμαστε τώρα, αν έχουμε για παράδειγμα παραδείγματα όπως το PNR, τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών ή άλλα, ή επίσης την εντολή εκτέλεσης έρευνας που υπάρχουν σε όλες τις αστυνομικές αρχές, αν περιληφθούν και αυτά, σε διαμεθοριακή ανταλλαγή, αυτά δεν μπορούν να κριθούν ξεχωριστά. Είναι σημαντικό λοιπόν να λεχθεί εδώ ότι η διακλάδωση, αυτή η διασύνδεση θα συνεχιστεί. Η συνεργασία των αστυνομικών αρχών και των δικανικών αρχών στην Ευρώπη θέλουμε αυτά να τα προωθήσουμε, αλλά χρειάζονται ενιαίες προδιαγραφές, ενιαία στάνταρ. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε πολύ ευαίσθητο ε, πεδίο εδώ, όπου υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ρυθμίσεις και γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι στην οδηγία μπορούμε να θεσπίσουμε μόνο ελάχιστε προδιαγραφέ, που όμω δεν μπορούν να έχουν αυθαίρετο χαρακτήρα και να αφήνουν τι υπόλοιπε ρυθμίσει τη ε, χώρε μέλη. Διότι όσο περισσότερο θέλουμε να διασυνδεθούν οι δραστηριότητε των διαφόρων αρχών, τόσο περισσότερο πρέπει να εναρμονιστούν αυτές οι ασφαλιστικές ρήτρες, οι safeguards. Δεν θέλουμε δηλαδή στο ευρωπαϊκό επίπεδο να λειτουργούμε ανεξαρτήτως από τα εθνικά επίπεδα και να φτιάχνουμε κάποιους οργανισμούς. Θέλουμε να διακλαδωθούν, να διασυνδεθούν οι εθνικές αρχές. Όποιος ωστόσο προωθεί αυτή τη διασύνδεση των εθνικών αρχών πρέπει ταυτόχρονα να καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες πρέπει όλο και περισσότερο και ακόμα περισσότερο δηλαδή να γίνουν ενιαίοι και άρα χρειάζεται και περισσότερη συγκεκριμενοποίηση, διότι σε πολλούς κανόνες αφήνεται μεγάλο περιθώριο για την εφαρμογή τους στις χώρες μέλη και είναι ασαφές ποιες είναι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που ισχύουν για την διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και, για παράδειγμα, σε θέματα όπως η διάρκεια αποθήκευσης παρά τις αρχές. Για παράδειγμα, δεδομένα PNR και άλλα. Όπου η οδηγία αυτή οφείλει να προβεί σε ευρύες ρυθμίσεις. Και ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι αυτό του λεγόμενου profiling. Γιατί η διασύνδεση διαφόρων τραπεζών δεδομένων έχει αρχίσει και γίνεται πια καθημερινή. Κάθε φορά που συζητούμε για χρήση δεδομένων και γι' αυτό χρειάζονται πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Και εγώ άλλωστε τάσομαι πάντοτε υπέρ της ιδέας να προσανατολιστούμε στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως άλλωστε κάναμε και εμείς στις διατυπώσεις που επιλέξαμε στις εκθέσεις μας. Και θα αρκεστώ σε αυτά. Θα αποταλθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο, να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που δίνετε να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Θα επικεντρώσω την προσοχή μου στον κανονισμό. The excellent uh, report. Εξετάσαμε την εξαιρετική έκθεση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Κομισιόν πάντοτε σώταν υπέρ της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών για την προστασία των δεδομένων. Α, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Τώρα συζητούμε την οδηγία, όχι τον κανονισμό. Μετά τον κανονισμό. Μετά. Α, τότε καλά. Για την οδηγία προς το παρόν θα περιοριστώ να πω ότι βεβαίως η Κομισιόν την πρότεινε ήδη μέσα στο πνεύμα της αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων των χωρών μελών. Γι' αυτό και είναι οδηγία και όχι κανονισμός. Γνωρίζουμε καλά την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες ε, της αστυνομικής δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και πρόοδος της δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων, παραδείγματο χάρη, για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Οποτεδήποτε παίρνετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα οπουδήποτε στην Ένωση βρίσκεται στην τράπεζα δεδομένων αυτήν. Ήδη υπάρχει αυτό και σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθεί το δίκτυο αυτό ανταλλαγής δεδομένων με κοινού κανόνες που να αυξάνουν κάπως το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με το πλαίσιο της οδηγίας και να εφαρμόζονται επίσης η προστασία αυτή και εθνικά για τα δακτυλικά. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ κάποια συνένεση που λέει να εφαρμοστούν τα ελάχιστα δυνατά πρότυπα και πολλές χώρες μέλη θα συμφωνούσαν από αυτού στο Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν έχει πρόβλημα με αυτό εφόσον αυτά τα ελάχιστα πρότυπα είναι επαρκώς επαρκή για να εξυπηρετούν το στόχο μας, δηλαδή την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτή την εποχή που υπάρχει τόσο αυξημένη δικτύωση. Ευχαριστούμε και τώρα πάλι το λόγο θα σας το δώσω αργότερα για τον κανονισμό. Τώρα ο κύριος Δρούτσας παρακαλώ για να καταλήξει. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα γερμανικά γιατί οι περισσότεροι σχολίασαν στη γλώσσα αυτή. Πολύ σύντομα τώρα για το ουσιώδες περιεχόμενο δεν θέλω να επισέλθω γιατί όλα τα σχόλια που ακούστηκαν είναι ιδιαίτερα ορθά και θα έχουμε και την ευκαιρία στη διάρκεια της διαδικασίας για τις τροπολογίες να συζητήσουμε εντατικά για τα θέματα αυτά. Τα όσα άκουσα από τις και τους αξιότιμους συναδέλφους μου εδώ σήμερα εντάσσονται στο πνεύμα της εκθέσεώς μου και προσωπικά είμαι πολύ ανοιχτός για να κατευθυνθώ προς την κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά ιδίω τι προτάσεις του Άξελ Βό, νομίζω δεν απέχουμε πολύ. Να προσθέσω κάτι γενικότερο μόνο. Στο θέμα που έθεσε ο κύριος Βος για την σύγκρουση αυτή που ασφαλώς δεν υπάρχει στο υλικό της οδηγίας, δηλαδή αφενός η προσπάθεια ενίσχυσης των δικαιωμάτων του ατόμου, από την άλλη μεριά η αποτελεσματικότητα της κρατικής ε, προσπάθειας αντιμετώπισης ενδεχομένων κινδύνων κλπ. Δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για σύγκρουση, διότι περισσότεροι έλεγχοι θα οδηγήσουν σε ε, αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων εφόσον προστατευτούν περισσότερο τα δικαιώματα του ατόμου, αυτό βρίσκω ότι είναι και ο καλύτερος και ο πιο σωστός δρόμος. Και το ερώτημα τώρα, ποιον στόχο θα πρέπει να επιδιώξει η οδηγία, περισσότερο μια εναρμόνιση ή περισσότερο ένα καθορισμό ελαχίστων προδιαγραφών. Εφόσον μιλούμε για ελάχιστε προδιαγραφέ, τότε θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με άλλου που μίλησαν προηγουμένω. Αν πρόκειται να μιλήσουμε για ελάχιστε προδιαγραφέ, αυτέ πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλέ. Ελάχιστε μεν υψηλέ δε. Ε, είμαι απολύτως εν γνώση και είμαι και ρεαλιστής. Γνωρίζω τα επιχειρήματα που ανέφερε ο Άξελ για τις διαφορετικές ε, νομικές παραδόσεις των χωρών μελών, ότι βεβαίως οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να επέλθουν προσεκτικά και βήμα-βήμα, όλα αυτά τα γνωρίζω. Από την άλλη μεριά και όπως είπα είμαι ρεαλιστής, δηλαδή εν τέλει θα έχουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, δηλαδή με τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να επιτύχουμε εν τέλει κάποιο αποτέλεσμα, πρέπει να βρούμε την απαραίτητη ισορροπία. Αυτό είναι απόλυτα σαφέ για μένα. Από την άλλη μεριά όμω, θέλω να τονίσω ότι εμεί εδώ, ιδίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να ερμηνεύσουμε σωστά και το πνεύμα των καιρών, για το μέλλον δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω αυτό και είμαι πεπισμένος ότι Εάν θέλουμε μια περαιτέρω ολοκλήρωση, μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πρέπει επιτέλους να τολμήσουμε να κάνουμε και το βήμα αυτό. Σε φακέλου, σε θέματα του πρώην τρίτου πυλώνα, όπου δηλαδή μπαίνουμε πια στο μεδούλι του κοκάλου των, ε, της αρμοδιότητας των κρατών μέλων. Θα χρειαστεί λοιπόν εν τέλει να γίνει μια προσπάθεια προς κάποια εναρμόνιση. Ευχαριστώ κύριε Δρούτσα. Τι ωραία ε, γερμανικά που μιλάτε, εκπληκτικό. Και ας προχωρήσουμε τώρα στον κανονισμό. Αυτό που είπα πριν, για την οδηγία τα ίδια ισχύουν εδώ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 27η Δευτέρου. Ας λάβει τώρα το λόγο ο κύριος Άλμπρεχτ, εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως συζητήσαμε και για την οδηγία, θα επανέλθω και εδώ στα όσα ήδη έχουμε συζητήσει στην πρώτη μας ε, συζήτηση. Δηλαδή, από πού ερχόμαστε, ας το πω έτσι, για να μιλήσουμε για τον κανονισμό αυτό. Ποιο είναι το αίτημα που έχουμε και που Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή το έχουμε ζητήσει και ξαναζητήσει και εν τέλει μάλιστα με το ψήφισμά μας του Ιουλίου 2011. Ότι δηλαδή από, την, ε, από τις εμπειρίες των τελευταίων 15 ετών με την παλαιά οδηγία διδαχτήκαμε ότι η διαφορετική εφαρμογή του δικαίου προστασίας δεδομένων στις χώρες μέλη έχει οδηγήσει σε εξασφάλιση της προστασίας αυτής σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες χώρες μέλη. Με αποτέλεσμα, από την άλλη μεριά, να υφίσταται μια σημαντική ανασφάλεια δικαίου και από την πλευρά των θυγωμένων αλλά και από την πλευρά των αρχών ή οργανισμών που χειρίζονται αυτά τα δεδομένα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε και μάλιστα σε απλουστευμένη βάση, δηλαδή χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει ένας ισχύων κανόνας που ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη και αυτός πρέπει να είναι. Όχι 27 διαφορετικές ενόμες τάξεις εν προκειμένου. Και αυτό είναι σημαντικό διότι χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση. Υπό την ισχύ της Παλαιά οδηγία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση. Εδώ, ωστόσο, πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος είναι κατεξοχήν διαμεθοριακός. Το 1995 το ίντερνετ δεν ήταν ακόμα μαζικό μέσο ενημέρωσης. Σήμερα ο καθένας είναι διαρκώς μέσα στα δίκτυα. Ανά πάσα στιγμή κάπου είμαστε συνδεμένοι με κάποιο δίκτυο. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για τους επιχειρηματίε και για τα άτομα, τους απλούς καταναλωτές και για τις αρχές. Γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να πω ως πρώτο ότι το επιδιωκόμενο είναι μια ενισχυμένη εναρμόνιση. Αυτό είναι ήδη σημαντική πρόκληση, διότι εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικές κουλτούρες προστασίας δεδομένων και για να φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Εφόσον πρόκειται για τον εντεταλμένο την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα σε μια επιχείρηση. Ήδη αυτό χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση. Και χρειάζεται και μεγάλη διάθεση συμβασμού από όλε τι πλευρέ. Και γι' αυτό νομίζω ότι ιδίω είναι σημαντικό από τη δική μα σκοπιά να καθιστούμε σαφώ διαρκώ ότι δεν θέλουμε κάτι το απολύτω νέο. Θέλουμε να βασίσουμε τη ρύθμιση αυτή στο δίκαιο και στην ομολογία που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και στις διάφορε χώρες μέλη, αλλά και διεθνώς. Έχουμε για παράδειγμα την Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην παραπέρα εξέλιξη προστασία δεδομένων στην Ευρώπη. Να ανατρέψουμε κάποιε υφιστάμενε βασικέ αρχέ. Και ο δρόμο που ακολουθήσαμε του τελευταίους μήνε ήταν να πούμε ότι οι ορισμοί και οι βασικέ αρχέ που έχουμε βάλει και στην οδηγία και στον κανονισμό ακολουθούν κατά βάση τις υφιστάμενες γραμμές. Μόνο που θέλουμε να οριστούν με ακριβέστερο τρόπο και θέλουμε εν τέλει κανονισμό που να είναι εφαρμόσιμος και εφαρμοστός και εφαρμοστέος για τον καθένα και την καθεμία από μας. Ένας στόχος που θα πρέπει να έχουμε διαρκώς υπόψη μας και όταν θα καταθέσουμε τροπολογίες. Σε πολλά από τα τμήματα που είχαμε ζητήσει με το ψήφισμά μας του Ιουλίου 2011, αυτά τα έχουμε λάβει ως βάση. Έχουμε τώρα άρθρα και ε, άρθρα της ιδεολογικής σκέψης, τα εκτιμώντας δηλαδή, με τα οποία και στον κανονισμό και στην οδηγία άλλωστε, που προσπαθούμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα στους επιμέρους τομείς και να πληρώσουμε όλα τα υφιστάμενα κενά. Και αυτό ήδη είναι ένα τεράστιο καθήκον. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στις τροποποιήσεις που επιφέραμε για μας, σημαντικό ήταν πρώτα να διαμορφωθούν οι ορισμοί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σαφές ότι τα όσα έχουμε λάβει από την ομολογία των τελευταίων ετών περνούν και στο κείμενο. Ιδίως για το προσωπικό δεδομένο, όχι είναι μια θεμελιώδης απόφαση το τι είναι προσωπικό δεδομένο. Γιατί αυτό θα κρίνει εάν θα ισχύει ο κανόνας στον χειρισμό ορισμένων δεδομένων. Και αυτό ισχύει για όλους τους ενδιαφερομένους, όπως είπα, πρόσωπα, επιχειρήσεις, αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί και ποιες νομικές επιπτώσεις θα προκληθούν. Επίσης, η μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ατόμου και οι υποχρεώσεις των χειριστών των δεδομένων, που να είναι σαφές ότι ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές, κάποια, δηλαδή κάποιους στόχους προστασίας, οι αρχές είναι αυτές που μας κατευθύνουν, σε αυτές προσανατολιζόμαστε και αυτές αντικατοπτρίζονται και στα δικαιώματα του καθενός ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, την ενημέρωση, την διαγραφή και την διόρθωση. Αυτά είναι σημαντικά δεδομένα τα οποία εξακολουθούν βεβαίως να υφίσταται και τα οποία έχουν και το αντίστοιχό τους σε ό,τι αφορά τις υποχρώσεις των αρχών που χειρίζονται τα δεδομένα και οι οποίες είναι υποχρεωμένε να προσφέρουν προστασία αλλά και ενημέρωση σε ό,τι είναι πράγματι απαραίτητο έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα επιμέρους δικαιώματα του ατόμου. Αυτό είναι το δεύτερο στο οποίο βασιστήκαμε και καταλήξαμε πάλι στο ότι για παράδειγμα η υποχρέωση ενημέρωσης περιορίζεται στα όσα είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο πρόσωπο για να μπορέσει να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Και επομένως και τα χορηγόμενα έγγραφα πρέπει να είναι αυτά που είναι απόλυτα απαραίτητα για τον χειριστή για να μπορεί να αποδεικνύει ότι έχει τηρήσει όλους τους κανόνες. Άρα, υποταγή στο εφιστάμενο δίκαιο. Ε, δεν πρόκειται και για πυρηνική φυσική εν τέλει, απλά πράγματα λέμε. Ότι θέλουμε να φτιάξουμε τους υφιστάμενους κανόνες έτσι που να είναι κατανοητοί. Η μεγάλη πρόκληση τώρα που συζητείται εντονότατα σε όλους τους κύκλους ενδιαφερομένων, τα λεγόμενα one-stop shop και το μηχανισμό συνεκτικότητας, δηλαδή ποιος είναι αρμόδιος για την ερμηνεία και την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων από την άποψη των αρχών χειρισμού. Ποιος είναι αρμόδιος και σε περίπτωση σύγκρουσης ποιος έχει τον τελευταίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή κατέστησε σαφέ αυτό που λέμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε την μοναδική αυτή θηρίδα, το One Stop Shop, να μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάθε χειριστής έχει έναν επιτετραμένο την προστασία προσωπικών δεδομένων με τον οποίο συνεργάζεται, που ο οποίος είναι αρμόδιος εάν κάτι δεν πάει καλά και εκεί ε, στην ε, δικαιοδοσία του οποίου γίνεται και η εκδίκαση των διαφορών. Επίσης όμως ο κάθε φυγόμενος μπορεί να απευθυνθεί στον δικό του επιτετραμένο προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λύση μεταξύ, στη συγκρούση δηλαδή μεταξύ αυτών των επιτετραμένων την προστασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε συνεργασία μεταξύ τους σε αναζήτηση κοινή λύση. Κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα και αποδίδει. Και μόνο εάν προκληθεί σύγκρουση, μόνο τότε καλείται η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πλέον να ασχοληθεί με το θέμα και θα έχει και τη δυνατότητα σε τελική φάση να λάβει απόφαση απόφαση την οποία θα καλείται να σεβαστεί ο επιτετραμένος στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Και σε απολύτως τελευταία φάση, με πλειοψηφία δύο τρίτων, η Επιτροπή αυτή μπορεί και να καταστήσει αναγκαστικώς εκτελεστή την αποφασή της. Πάντως, αυτή ήταν η, η πρόθεσή μας, να καταστήσουμε σαφές δηλαδή ότι αυτό είναι το επιθυμητό από εμάς και ότι δεν είναι εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη η οποία θα καλείται να κρίνει επί της αποφάσεως ενός επιτετραμένου. Αλλά θα είναι σαφές ότι αν αυτό έχει κρίνει ο επιτετραμένος, τότε πλέον είτε τα δικαστήρια είτε ο νομοθέτης, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα κληθούν να κρίνουν αν απαραίτητο ας πούμε να υπάρξει μια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου ή όχι. Είναι και συμβατικά εξασφαλισμένη η αρμοδιότητα των επιτετραμένων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα, διότι αφενό είναι σαφέ ότι μόνο ο νομοθέτης μπορεί να θεσπίσει δίκαιο και αυτό το βάζουμε και στον κανονισμό. Και γι' αυτό και διαγράφουμε πολλές και εκτελεστικέ πράξει και τι αντικαθιστούμε με ορισμένε διακριβώσει μέσα στο κείμενο. Από την άλλη μεριά είναι σαφέ ότι και οι επιτραμένοι την προστασία των δεδομένων πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το σχετικό δίκαιο. Και αυτό βέβαια χέρι διαφόρων ερμιών. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Ασφαλώς θα το συζητήσουμε κι άλλο. Πάντως είναι σαφές ότι αυτό που θέλουμε είναι ενία, μάλλον εξασφάλιση της ενία εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό πρέπει να είναι ο απότατο στόχος μας, διότι όπως είπα και στην αρχή αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ασφάλεια δικαίου με τον κανονισμό που θεσπίζουμε αλλά και με έναν μηχανισμό συνοχής που θα εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή. Όπως είπα χαίρομαι ιδιαίτερα που θα υποβληθούν και τροπολογίες οι οποίες ασφαλώς θα βελτιώσουν το κείμενο. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε και με τους σκιώδεις εισηγητάς και να προσπαθούμε κατά το δυνατό όλο αυτό το περίπλοκο υλικό να σας το υποβάλουμε με μια μορφή που να είναι δυνατό να ψηφιστεί εν τέλει. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και η προσωπική μου παράκληση, αλλά νομίζω και των άλλων συναρμοδιών, είναι να ρίξετε το βάρος σας ιδίω σε εκείνα που πραγματικά είναι σημαντικά και που πρέπει να τροποποιηθούν, διότι πολλά τα έχουμε ήδη συζητήσει πριν να επιφέρουμε τις τροποποίησεις αυτές. Εάν λοιπόν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες, ξανασυζητήστε, με τους και τις των ομάδων σας, διότι εν τέλει το κείμενο πάει να γίνει τόσο περίπλοκο και σίγουρα θα υποβληθούν τόσες πολλές τροπολογίες, ώστε στο τέλος θα είναι μακροτάτη η διαδικασία ψηφοφορίας. Και για να απλουστεύσουμε λίγο τη ζωή μας, καλό είναι η πρώτερη καλή συνεργασία, διότι θέλουμε να προχωρήσουμε και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, πριν επομένω από τον επόμενο προεκλογικό αγώνα. Έρχομαι αμέσω σε αυτά που είπε και ο Σάλμπεχτ. Πράγματι, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητούμε για να γίνονται σχετικές βελτιώσεις. Σωστό επίσης είναι ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η ενιαία εφαρμογή του όλου αυτού, του συνόλου των ε, κανόνων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλαίσιο για την προστασία δεδομένων που θα λαμβάνει υπόψη μια ανάγκη εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το άτομο αλλά και επιτρέποντάς του επαρκές περιθώριο ελευθερίας και έκφραση και ανάπτυξη προσωπικότητά του. Δηλαδή, εάν φτάσουμε σε κάποια ακραία όρια προστασία των δεδομένων, σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κινηθεί το πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και πώς, ποια είναι η αλληλεπίδραση των διαφόρων κανόνων. Ο πολίτης αφενός θέλει να είναι προστατευμένος, η προσωπική του σφαίρα, τα δεδομένα του, ταυτόχρονα όμως επιθυμεί να μπορεί να εκμεταλλεύεται προσφορές που για παράδειγμα φέρνω παράδειγμα ε, προσφορές δωρεάν στο διαδίκτυο. Εάν αν υπερβάλλουμε την προστασία αυτή τότε ενδέχεται να μην μπορεί να δει αυτές τις προσφορές ή να μην μπορεί να τις πληρώσει. Αυτά τα είχα πει και την προηγούμενη φορά. Και ενδεχομένως ε, με την υπερβολική προστασία να φτάσουμε και σε πολύ αυξημένες τιμές τέτοιων προσφορών. Και τότε δεν προσφέρουμε καμιά μεγάλη υπηρεσία στον πολίτη. Άρα χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία των συμφερόντων του ατόμου, να έχει δηλαδή προστατευμένα τα δικαιώματά του, αλλά ταυτόχρονα να έχει και ένα περιθώριο ανάπτυξη προσωπικότητά του. Και εδώ νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο. Ελευθερία, αυτοδιάθεση, αυτοευθύνη, όλα αυτά είναι και για μας και σημαντικές πηξίδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό τον μηχανισμό συνοχής ή συνεκτικότητας που ανέφερε ο κ. Άλμπρεχτ και που εξήγησε τι εννοεί και πόσο σημαντικό είναι για να φτάσουμε στην ενιαία εφαρμογή και να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσέγγιση του One Stop Shop είναι απόλυτα σωστή και λογική και μπορεί να οδηγήσει στα ανάλογα αποτελέσματα. Κάτι που βρίσκω να λείπει, ωστόσο, είναι ένα είδος διορθωτικού μηχανισμού. Δηλαδή, αν έχουμε, αν αφήσουμε μονάχα στο, στο μηχανισμό προστασίας των δεδομένων την ευκαιρία να λύνει τα προβλήματα, τότε αυτό θα γίνεται στη βάση της προστασίας. Στους, στις προβληματικές όμως περιπτώσεις ίσως να μην λαμβάνονται υπόψη άλλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία χρειάζεται να εξισορροπηθούν. Αυτή την εξισορρόπηση πρέπει κάπω να την εξασφαλίσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι θα έλεγα ότι δεν πρέπει να αφήσουμε σε άλλου να κάνουν τη δική μα δουλειά. Εμεί είμαστε ο Ευρωπαίος νομοθέτης και σε περιπτώσει διαφορών πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, διότι αλλιώ διατρέχουμε τον κίνδυνο είτε η διοίκηση είτε η επι, την προστασία των δεδομένων να υπησέλθουν στο δικό μας ρόλο. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο, το γνωρίζω. Γι' αυτό η προσέγγιση του Γιάνν Φίλιπ είναι λογική. Όμως, ακόμα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει πετύχει την απαραίτητη ισορροπία που επιθυμώ να δω εγώ ως νομοθέτης. Πρέπει να αναρωτηθούμε επίσης και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον προβληματισμό του λεγόμενου direct marketing. Πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο εδώ, να δούμε αυτά τα μέτρα, τι επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν. Εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Και νομίζω ότι εδώ στην πρόταση του εισηγητού αυτά δεν έχουν ληφθεί ακόμα απολύτως υπόψη. Ώστε και εδώ χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Ένα άλλο θέμα είναι, και πολλοί το βλέπουν αυτό κάπως αρνητικά, είναι αυτό το λεγόμενο profiling. Έχουμε έναν ευρύτατο ορισμό για την ώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις αλλά και τις διασυνδέσεις. Δηλαδή ακόμα και μια επιχείρηση η οποία επιθυμεί να επικοινωνήσει με όλους τους πελάτες της, αλλά ίσως θέλει να κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε πελάτες πρώτης κατηγορίας συντοσιακών και δεύτερης, ενδέχεται να υπάρξει και εκεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή τότε δεν μπορεί πια η επιχείρηση να δράσει με τον τρόπο που επιθυμεί και που είναι λογικός. Εδώ λοιπόν βρίσκω ότι αυτός ο ορισμός είναι υπερβολικά ευρύς. Και εδώ χρειάζεται να βρούμε μια πιο ρεαλιστική λύση. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης, εδώ πρέπει να εξεταστεί εάν ίσως χρειάζεται κάποιο όριο στην περίπτωση που ενδέχεται να υπάρξουν καταχρήσεις. Εάν δηλαδή κάποιος σε μηνιαία βάση έρχεται και ζητά ενημέρωση για το φάκελό του. Ε, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαρκώς, ας πούμε σε μηνιαία βάση όπως είπα. Ίσως είναι υπερβολικό. Και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε αν αυτό καλύπτεται ή όχι. Για το λεγόμενο δικαίωμα να ξεχαστείς, right to be forgotten. Εκεί πρέπει να επιδιώξουμε μια τεχνικά εφαρμόσιμη λύση. Και αυτό εν μέρει έχει γίνει. Αλλά να δούμε ότι αυτό δεν μπορεί παρά μόνο οικειοθελώς δηλωμένα δεδομένα. Και τώρα για την Data Bridge Notification εκεί πρέπει να συζητήσουμε αν θα περιοριστούμε στο χρονικό προσδιορισμό που περιλαμβάνεται εδώ ή εάν θα εξετάσουμε περισσότερο την βαρύτητα των παραβιάσεων της ε, προστασίας των δεδομένων. Αυτό που βρίσκω σωστό είναι η αυτορύθμιση για τις επιχειρήσεις και ιδίω σε ό,τι αφορά τον επιτετραμένο προστασία δεδομένων της επιχείρησης και κάτω από τη σκοπιά της διαφάνειας που εδώ πρέπει να τονιστεί πράγματι ο ρόλος του. Εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν και έχουμε και ορισμένα άλλα θέματα για παράδειγμα τον ορισμό του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν δούμε τώρα αναφορικά με την διατύπωση το λεγόμενο singling out το θεμητό συμφέρον ή το νόμιμο συμφέρον να δούμε αν όντω δηλαδή έχουμε επιτύχει όλα αυτά Άλλε μορφέ δεδομένων είναι και εδώ σημαντικέ, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ ναι μεν η προσέγγιση είναι σωστή, αλλά δεν προχωρούμε αρκετά, ενώ τα ψευδονυμικά δεδομένα για να δίνονται δηλαδή στις επιχειρήσεις. Ας αρκεστώ σε αυτά και θα έχουμε τη δυνατότητα και στην ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών να εγκύψουμε σε λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις αυτές. Αλλά ακόμα θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στην αντιστάθμιση αυτή που χρειαζόμαστε για την προστασία του πολίτη σε αυτή την διοικότητά του, δηλαδή αφενός προστασία, των, ε, ε, προστασία της προσωπικής του σφαίρας αφενός αλλά και ταυτόχρονα ένα περιθώριο για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη. Η κυρία Ζίπελ. Επανέρχομαι στα όσα είπε ο κύριος Άλμπρεχτ στην αρχή, δηλαδή ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά βασιζόμαστε σε υφιστάμενα θεμέλια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι υπάρχουν πολλοί φορείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ λογικά την πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν και άλλοι όμως που προσπαθούν να προκαλέσουν την εντύπωση στην δημόσια αυτή συζήτηση που γίνεται σαν δήθεν να δημιουργούμε νέα πολύ αυστηρά νομοθετήματα. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένοι που θεωρούν ότι που μάλλον πάνε να φτιάξουν να προτείνουν και άλλες, και άλλες έξτρα προστασίες ώστε μετά να πούν ότι όλα αυτά δεν είναι ρεαλιστικά. Θα έρχω σε λίγα από τα θέματα που έφυξε ο κύριος Βος, ε, ε, επί των οποίων διαφωνώ. Βεβαίως πολλοί χρησιμοποιούν ιδίω για τα ηλεκτρονικά μίδια προσφορές που είναι δωρεάν. Όμως δεν γνωρίζουν όλοι ποιο είναι πραγματικά το τίμημα αυτών των δωρεάν προσφορών. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Εάν παραγγέλνω τακτικά βιβλία αλλά και ορισμένα καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα. Είναι γνωστό αυτό και μπορεί όντω να δοθούν τα δεδομένα αυτά και σε δύο-τρει άλλε εταιρείε παραπέρα. Άλλοι πολίτε μπορεί να πούν, εγώ δεν το θέλω αυτό, άλλοι πολίτε όμω μπορούν να πούν, «Ε, ναι, εμένα μου αρέσει πολύ να δώσετε τα δεδομένα μου και παραπέρα σε άλλε εταιρείε, γιατί τότε ίσω να μου υποβάλουν και άλλε ενδιαφέρουσε δωρεάν προσφορέ. Αυτό όμω πρέπει να το κρίνει ο κάθε ένα ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, όμω, όπω είναι τώρα τα πράγματα δηλαδή, δεν γνωρίζουμε καν εάν διατίθεται περαιτέρω τα δεδομένα. Επομένως, εκεί χρειάζεται προστασία. Ακόμα, τα δεδομένα μετακινούνται εσωτερικά σε μια επιχείρηση από αυτήν η οποία αποστέλει τα βιβλία σε άλλο τμήμα της ίδιας επιχειρήσης η οποία για παράδειγμα κάνει προσφορές για ταξίδια. Το πρόβλημα τώρα ότι ορισμένα δεδομένα ή ορισμένες προσφορές υπηρεσιών δεν θα είναι πλέον, στην περίπτωση αυτή που εξήγησε ο κ. Βος, δωρεάν. Εγώ δεν βρίσκω να είναι πρόβλημα αυτό με την έννοια ότι κάτι θα πρέπει να προστατευτεί. Για παράδειγμα, το ίδιο είναι το κατέβασμα δωρεάν βιβλίων ή ταινιών, που συχνά όμως είναι παράνομα. Είναι καλύτερα να πάει κανείς να ε, λάβει για παράδειγμα προσφορές πολύ φθηνές για το κατέβασμα βιβλίων ή ταινιών που εξακολουθούν όμως να είναι πολύ πιο συμφέροντα από το να πάει να τα αγοράσει έξω στο εμπόριο. Όλα αυτά δεν είναι δωρεάν γιατί ο καταναλωτής τα πληρώνει με τα δεδομένα του. Πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να έχει δυνατότητα να πει όχι, εγώ προτιμώ να πληρώνω μια μηνία συνδρομή και να μην μεταφέρω τα δεδομένα μου παραπέρα. Τώρα, υπάρχουν πολλές λύσεις για το direct marketing, πολλές εφημερίδες λένε ότι εάν ο, ο καταναλωτής πρέπει κάθε φορά να δέχεται ρητά την παραπέρα μετάδοση των δεδομένων του, τότε οι επιχειρήσεις αυτές λένε ότι θα καταστραφούν. Ναι, αλλά άμα πάω εγώ στον ε, ράφτη και του παραγγέλνω σακάκια κάθε τόσο. Δεν θέλω απαραίτητα να δώσει αυτό στη διεύθυνσή μου και το όνομά μου σε μια επιχείρηση κυπουρική που να μου στέλνει μετά προσφορέ για έπιπλα κήπου. Επειδή θεωρεί ότι ίσω εγώ έχω το ενδιαφέρον αυτό. Άλλωστε πολλά από αυτά καταλήγουν και στα σκουπίδια. Κάτι άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ο φόβος εκείνος ότι πρέπει να περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβαση στην ενημέρωση, επειδή λέει κάποιος μπορεί να ρωτάει τρεις φορές την εβδομάδα κάποιον πάροχο υπηρεσιών, μα ποια δεδομένα έχετε δικά μου στη διάθεσή σας. Μα αυτό ενδέχεται να περιορίσει εκείνους οι οποίοι ούτως ή άλλως κάποτε κάπου κάπου ζητούν να μάθουν ποια ε, προσωπικά δεδομένα έχουν αποθηκευτεί. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι υπερβολικά λίγες οι πληροφορίες και ότι υπερβολικά λίγοι πολίτες ζητούν να μάθουν ποιος διαθέτει τα δεδομένα τους και για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιεί. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να βάλουμε και άλλα εμπόδια στους πολίτες. Ούτως ή άλλως είναι συχνά δύσκολο σε θέματα δικαιώματος αντίθεσης ή εάν για παράδειγμα δεν θέλω ένας ε, πάροχος υπηρεσιών να διαθέτει ε, τα δεδομένα μου ή θέλω να του ζητήσω να τα διαγράψει, δεν βρισκό ποιος είναι ο συνομιλητής μου. Ή, για παράδειγμα, μπορώ μεν να, ε, να, κάνω, να υποβάλω παραγγελίες επιγραμμικά με το ίντερνετ, αλλά για να διταχθώ στην παραπέρα χρήση των δεδομένων πρέπει να στείλω γραπτή επιστολή. Δηλαδή γίνεται πιο δύσκολο. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφέ ποια πράγματα επιτρέπονται και ποια δεν επιτρέπονται και επίσης ποια πράγματα πρέπει να αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια των πολιτών. Και για όλους τους ενδιαφερομένους εν τέλει είναι σημαντικό, άλλωστε αυτό υπήρξε και αφορμή για να συνταχθεί το νέο κείμενο, οι αρχές της προστασία δεδομένων, δηλαδή οι βασικέ αρχέ, να μπουν σε μια νέα ευρύτερη βάση, έτσι ώστε και οι επιχειρήσει στο μέλλον να μην ψάχνουν να βρουν έδρες όπου η έλεγχη να είναι πιο χαλαρή, αλλά να υπάρχουν κοινά επίπεδα προστασίας σε όλες τις χώρες. Ίσως κάποιοι επικρίνουν ότι η προστασία αυτή που προτείνουμε είναι υπερβολική, αλλά μην λησμονούμε ότι δεν πρέπει να πέσουμε θύμα εκείνων οι οποίοι τα βλέπουν όλα μαύρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάντφορντ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που έχω χάσει τη φωνή μου. Δεν είμαι εισηγήτρια, αλλά θέλω να σχολιάσω ένα συγκεκριμένο θέμα για το οποίο μου μίλησαν πολλοί ακαδημαϊκοί. Τη σχέση δηλαδή του άρθρου 9, αν δεν απατώμε, με τα 80 και 83 όπου προτείνονται μάλιστα τροπολογίες και όπως σας είπα μου μίλησαν πολλοί ότι ανησυχούν για τη δυνατότητα αυτή μείωση της ακαδημαϊκής έρευνας με βάση θρησκευτικές ή πολιτικές πεπιθήσεις Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πόλεμος στο Ιράκ ή τα βασανιστήρια όπου μπορεί να υπάρχουν θεμητά, θεμητός σχολιασμός πολιτικός. Εμείς θέλουμε να γίνεται σεβαστό το δίκαιο πάντοτε και θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι ανησυχίες που μου εκφράστηκαν είναι λογικές ας πούμε. Η τροπολογία 336 το ότι τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να τα χειρίζονται για έρευνα μόνο με την άδεια του ενδιαφερόμενου. Σε πολλές περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος δεν θα ήθελε να γίνονται γνωστές οι απόψεις του ή η συμπεριφορά του με τρόπο που θα μπορούσε να τον σύρει στα δικαστήρια παραδείγματο χάρη. Και δεν είμαι βέβαιη σε τι βαθμό οι διατάξεις όπου στην τροπολογία 3-2-4 διευρύνεται η εξαίρεση από την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων γιατί λέει εκεί ότι οι εξαιρέσεις θα χορηγούνται οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για να συνδυαστεί η ελευθερία της έκφρασης με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καλό μένει είναι αυτό, αλλά αν δούμε μετά το 83 ή το 80 μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πώς οι ερευνητές θεμητοί, οι κανονικοί ερευνητές και ερευνήτριες. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε σταμα... που σταματάει η δημοσιογραφία και που αρχίζει η έρευνα, αλλά για θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος ξέρουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι ποτέ δεν θα έδιναν την άδειά τους για δημοσίευση τουλάχιστον. Θα το ξαναδώ λοιπόν από ό,τι ξέρω ο εισηγητής δεν θέλει πράγματι να μειωθούν οι έρευνες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να τα εξισορροπήσουμε όλα γιατί δεν θέλουμε να ανοίξουμε το κουτί της ανδόρας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν θα ήταν σωστό να καταλήξουμε να κλειδώσουμε την έρευνα ή τον την ερευνητική δημοσιογραφία. Αν και μπορεί πάντοτε ο ενδιαφερόμενος να μην έχει συμφέρον να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Θα το ξαναδώ λοιπόν. Ίσως να καταθέσω και άλλες τροπολογίες μάλιστα. Ευχαριστούμε και τώρα η Κομισιόν. Σας κατευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα υπενθυμίσω ότι για μας το Συμβούλιο στο Δουβλίνο την περασμένη Παρασκευή έκανε μια, διεξήγαγε μια καλή συζήτηση τις εξαιρέσεις για τα νοικοκυριά, τις διοικητικές κυρώσεις τυρκές κυρώσεις, και το δικαίωμα λύθης. Γενικά υποστηρίχθηκαν οι προτάσεις μας και βέβαια θα τις επεξεργαστούμε κι άλλο με το Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη για να υπάρξει περισσότερη συνένεση και να έρθουν όλα αυτά σε πιο νομική μορφή. Θα ήθελα τώρα να σας πω μερικά λόγια για τον μηχανισμό συνέπειας στους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Είναι βασικό αυτό, καθώς και το στοιχείο καινοτομίας που έχει ο κανονισμός ως προς την οδηγία. Καταρχήν η Κομισιόν πάλεψε και με το δικαστήριο για την ανεξαρτησία των αρχών που θα εποπτεύουν τα προσωπικά στοιχεία. Δεν έχουμε λοιπόν καθόλου την πρόθεση να υπονομεύσουμε την ανεξαρτησία των αρχών, εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων. Η ανεξαρτησία τους αναφέρεται ρητά στη συνθήκη. Τόσο ρητά που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο τμήμα των συνθήκων τέτοια σαφήνεια. Για μας είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι οι μηχανισμοί που λέγονται peer review και που αφορούν μόνο τις χώρες μέλη δεν συνδυάζονται πολύ καλά στην Ένωση. Οι μηχανισμοί που υπάρχουν όμως όπως την νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, την οδηγία της τηλεπικοινωνίας για τα σλότ των ε, αερομεταφορών συνεργάζονται οι εθνικές αρχές με κάποιο, κάποια διάσταση όμως και ενωσιακή συμμετοχή. Σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς δηλαδή η Κομισιόν παίζει τον νενομισμένο της ρόλο από τις συνθήκες, δηλαδή είναι θεματοφύλαξ του κοινού ενωσιακού συμφέροντος. Και γι' αυτόν τον λόγο προτείναμε ε, και έναν μηχανισμό που δεν επιτρέπει στην Κομισιόν να ανατρέψει αποφάσεις των εθνικών αυτών αρχών. Τους, τις επιτρέπει μόνο να παίζει το ρόλο που προβλέπεται να παίζει από τη συνθήκη και σε όλους τους μηχανισμούς όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών, δηλαδή εκπροσώπηση του κοινού συμφέροντος και διασφάλισης μιας εξισορρόπησης των διαφορετικών συμφερόντων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γενικά της κοινή αγοράς. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον είναι θεμητό και νόμιμο αυτό που προτείνεται εδώ. Μάλιστα συμμεριζόμαστε την άποψη των εισηγητών και άλλων που είπαν ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτά που ήδη υπάρχουν, όχι δηλαδή μόνο την παράδοση προστασίας των δεδομένων, αλλά και το κεκτημένο της ε, ενωσιακής νομοθεσίας. Εδώ έχουμε συνθήκη, η οποία κατόπιν ετοιμάτων του Κοινοβουλίου στο 190, στο άρθρο 190 και 191, χορηγεί δικαιοδοσίες στην Κομισιόν και αυτό με αίτημα κατόπιν αιτήματο του Κοινοβουλίου, το οποίο παίζει κάποιο ρόλο. Στι τροπολογίε όμως βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα παίζει πια κανένα ρόλο στην εφαρμογή δεσμευτικών κανόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Θα μας εξέπληξε το Κοινοβούλιο να ζητάει να μην υπάρχει ενωσιακή εκπροσώπηση πλέον του κοινού συμφέροντος. Τόσο για τις μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν στο δευτερογενές δίκαιο να δημιουργηθεί ένα σώμα εθνικών αρχών που να έχει το δικαίωμα να παίρνει δεσμευτικές αποφάσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο προτείναμε μηχανισμό που να καθοδηγεί και να δίνει στην Κομισιόν τη δυνατότητα μέσα σε ορισμένα όρια να κυρώνει ορισμένες μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά που τελικά θα αφήνει την ατομική απόφαση, τη μεμονωμένη απόφαση στις εθνικές αρχές. Και γιατί προτείναμε αυτή τη δυνατότητα ακύρωσης, για να δοθεί περισσότερος χρόνος αναλογισμού του τι είναι, σε τι συνίσταται, το κοινό συμφέρον. Καλούμε λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής σας να συνεργαστούν μαζί μας ώστε να βασιστούμε στις, εμπειρίες, στις θετικές εμπειρίες και άλλων ενωσιακών μηχανισμών συνεργασίας εθνικών αρχών με την Κομισιόν ώστε να διατηρηθεί αυτό το στοιχείο του κοινού συμφέροντος που εκπροσωπεί η Κομισιόν και σε αυτό το θέμα των μεμονωμένων λήψεων αποφάσεων. Τέλος επιθυμίζω επίσης ότι στην πρότασή μας άρθρο 66.1β το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει τη δυνατότητα να απευθύνει συμβουλές και ευέλτιστες εμπειρίες στα κράτη-μέλη, αλλά λόγω της ίδιας του της φύσης δεν είναι δεσμευτικές αυτές. Επίσης πρέπει να πω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι αν εργαστεί καλά αυτός ο μηχανισμός που βασίζεται στο, άρθρο 29 για την ερμηνεία των οδηγιών. Εάν ο μηχανισμός αυτός εργαστεί καλά, λειτουργήσει καλά μάλλον, τότε δεν θα υπάρξουν και τόσο πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις που να πρέπει να αποφασίζει. Διότι θα υπάρχει σαφήνεια εξάντε. Και αυτό χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να υπάρχει σαφήνεια πριν τεθεί συγκεκριμένο πρόβλημα και ταυτόχρονα εάν λειτουργήσει καλά ο μηχανισμός αυτός τότε μπορεί να μην υπάρξει και καμία ανάγκη για περισσότερη νομοθεσία σύμφωνα με αυτά που προτείνει το 190 και 191. Τώρα, σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός αυτός. Δεν χρειάζεται περισσότερη εξουσιοδότηση τη Κομισιόν για συνεργασία με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο όπως βλέπετε στι συνθήκε. Νομίζουμε ότι θα ήταν λάθο κάτι τέτοιο. Γιατί η πιθανότητα το σύστημα να, εργα... να λειτουργήσει καλά αυξάνεται αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ότι άμα δεν λειτουργήσει άμα κάποια εθνική αρχή δεν συμφωνήσει με τους κανόνες τότε μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν δεσμευτικοί κανόνες με, με τη μορφή you to uh, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Άρα μπορεί κανείς να πει ότι αυτές οι εξουσιοδοτήσεις για ό,τι είναι βασικό πρέπει να αποφασίζονται από τον ίδιο τον νομοθέτη. Τώρα όμως προτείνουμε, αυτό που προτείνουμε σημαίνει ότι όλη η εφαρμογή αφήνεται στα χέρια του σώματος που δεν προβλέπεται στον ενωσιακό νόμο και που δεν θα λειτουργούσε και σύμφωνα με τις εγγυήσει που σας δίνει στο 190 και 191 η συνθήκη να παίξετε και εσείς κάποιο ρόλο δηλαδή στην εφαρμογή της οδηγίας. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε το κοινό συμφέρον που εκπροσωπεί η Κομισιόν και ότι αυτό θα διατηρηθεί και στους μηχανισμούς αυτούς και στις μνημονικές επιπτώσεις και στις κατεξουσιοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλες και όλους τους συναδέλφους που ε, παρενέβησαν και δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο νόημα να επανέλθω σε όλα τα σχόλια που κάνατε. Άλλωστε τα θέματα θα τα συζητήσουμε εντατικά περαιτέρω. Και ίσως είναι καλύτερα να περιοριστώ σε μερικές γενικές παρατηρήσεις. Και πρώτα, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια και το κείμενο της Κομισιόν και τα δικά μας. Διότι ήδη μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται πάρα πολλέ σκέψεις και προβληματισμοί. Αυτά που εξήγησε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Consistency Mechanism. Υπάρχει και η δυνατότητα να εξεταστούν διαφορετικές οπτικές και δικό μου αίτημα είναι να διαβάσουμε όλοι προσεκτικά τις προτάσεις. Πολλές από τις παρατηρήσεις που γίνονται τώρα για τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει περιλαμβάνονται στα κείμενά μας. Ορισμένες φορές δεν είναι ίσως τόσο εύκολο να τις βρει κανείς. Για παράδειγμα, για τα ψευδόνυμα και για ορισμένα προσωπικά δεδομένα και που σωστά συζητούνται πολύ αυτά. Αν θα περιληφθούν κάπου ξεχωριστά. Για τα προσωπικά δεδομένα βασισμένα σε ψευδόνυμα, ωστόσο αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Το ίδιο το singling out, που σύμφωνα με τη μέχρι τώρα νομολογία και με τους ορισμούς που έχουμε, πάντοτε όταν μπορούσε να γίνει μια ταυτοποίηση τότε πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Και με την χρήση των ε, ψευδόνιμων ε, των δεδομένων Ναι, μεν δεν μπορεί να επιτευχθεί ταυτοποίηση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η ενδεχόμενη δυνατότητα ταυτοποίησης του προσώπου μέσω ορισμένων άλλων παραμέτρων των δεδομένων, έστω και με ψευδόνυμο. Έτσι λοιπόν, τα ψευδόνυμα δεδομένα είναι ένα τμήμα των προσωπικών δεδομένων που χρήζουν προστασίας. Επειδή τώρα προβαίνουμε στους ορισμούς αυτούς, κάνουμε τους ορισμούς αυτούς, βλέπουμε και μερικές εξελίξεις τώρα ιδίως στο online. Για παράδειγμα, αν βάλει κανείς, αν ε, βάλει ορισμένες ρυθμίσεις το browser που χρησιμοποιεί να μπορεί να αποφύγει την συλλογή των δεδομένων του. Αυτό είναι μια πιθανή οδός που μπορεί να εξεταστεί. Θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο απλή την χορήγηση της έγκρισης από πλευράς του προσώπου για την χρήση, για τη συλλογή δηλαδή και χρήση των δεδομένων του. Όμως είπε και η κυρία Ζήπελα άλλωστε αυτό μπορεί να είναι δυνατόν μόνο όταν το πρόσωπο μπορεί να χωρίσει την έγκρισή του, αλλά τελών ενήμερο του τι πράττει. Ο κανόνας λοιπόν πρέπει να είναι, όπως είναι τώρα, ο κανόνας είναι η έγκριση και η εξαίρεση μόνο είναι η μη χορήγηση της έγκρισης για την συλλογική χρήση των δεδομένων. Ενδεχομένω θα υπάρξουν κάποιες εξαιρεσει στις ρυθμίσει αυτές, αλλά ε, καλό είναι να ανοιχτούν τα χαρτιά, να μπορούν οι καταναλωτές να χορηγούν την έγκρισή τους, να μην τους προκαλείται η εντύπωση ότι ό,τι και να κάνουν είναι περιττό και στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις και ούτω καθεξής κάνουν ό,τι θέλουν. Μία σύντομη παρατήρηση, γιατί βλέπω ότι η κυρία λάντφορντ απεχώρησε ήδη, αλλά θα επανέλθω γιατί ίσως ενδιαφέρει άλλους. Οι ιδιαίτεροι κανόνες για την έρευνα και ιδίω όπου αυτή διεξάγεται και προς το κοινό συμφέρον, προς το δημόσιο συμφέρον. Είναι εκεί ιδιαίτερα δύσκολο να θεσπιστούν κανόνες. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να συγκεκριμοποιηθούν τα όσα είναι δυνατά στον τομέα της ε, έρευνας και για τον χειρισμό των δεδομένων εκεί αποκλείεται η στατιστική συλλογή ανωνυμοποιημένων δεδομένων δηλαδή συλλογή δεδομένων χωρίς ε, ταυτοποίηση του προσώπου είναι δυνατή. Αλλιώς υπάρχει ιδιαίτερη αναγκαιότητα, ιδίως για ευαίσθητα δεδομένα, Οι επιφυλάξει επιφυλάξεις της κυρίας Ντάτφορτ, ιδίω για την ελευθερία έκφρασης και νομικών διαδικασιών, αυτά εκπίπτουν με την έννοια ότι η ελευθερία έκφρασης, βλέπε άρθρο 80, είναι μια ιδιαίτερη έκφραση των προσωπικών της, προσωπική της ε, προσωπικής η οποία προστατεύεται από τα δικαστήρια και βεβαίως και από τους εθνικούς νομοθέτες οι οποίοι θεσπίζουν τους κανόνες για την ελευθερία έκφρασης. Ασφαλώς μπορεί να συζητηθεί αυτό, εάν δηλαδή μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι που μας απασχόλησε πριν εδώ πάλι στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και αν πρέπει να ρυθμιστεί αυστηρότερα ή αν πρέπει να υπάρξουν κοινοί κανόνες. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε βέβαια μέσα στον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, γιατί τότε δεν μπορούμε, δεν, το, κείμενο θα είναι ατελείωτο. Πρέπει να γίνουν εκ παραλλήλου Και σε ό,τι αφορά τι νομικέ διαδικασίε, είναι σαφέ ότι εφόσον κάτι ρυθμίζεται νομικά, εφόσον η έρευνα και η συλλογή στατιστικών δεδομένων θεσπίζονται νομικά, ρυθμίζονται νομικά, τότε αυτά καθίστανται δυνατά μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής. Αυτά ήθελα να συμπληρώσω και για τα υπόλοιπα είμαι ανοιχτός σε περαιτέρω συζητήσεις, άλλωστε χαίρομαι που θα γίνουν αυτές γιατί θα κάνουμε και μερικές συζητήσεις και μέσα στο Μάρτιο όταν θα έχουμε όλες τις τροπολογίες και όταν θα έχουμε και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα είναι σημαντικές για μας. Το ίδιο τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχολήσεως. Ευχαριστώ. Και πάλι προθεσμία για την υποβολή των ομολογικών 27 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Και πάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης για σήμερα το απόγευμα θα εξετάσουμε ένα έγγραφο εργασία, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια τη επικείμενη έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρότυπα και πρακτικέ στην Ουγγαρία. Το σχετικό έγγραφο θα μας το παρουσιάσουν οι δύο συντάκτες, ο κύριος Ταβάρες, ε, εισηγητής της έκθεσης και η κυρία Ρίπε. Πρώτα απ' όλα το λόγο έχει ο κύριος Ταβάρες και η κυρία Ρίπε έπειτα. Κύριε Ταβάρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνουν τώρα και γρήγορα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ένα λεπτό. Okay, thank you. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρίστανται σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το τρίτο έγγραφο εργασίας Όπω όπως είπαμε την αρχή συντάσσουμε με βάση το ψήφισμα του περασμένου Φεβρουαρίου και την επικείμενη έκθεση που πρέπει να εκπονήσουμε για θέματα δημοκρασίας, κρατός δικαίου, πολυφωνίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στην Ουγγαρία. Θα γνωρίζετε ότι βασικές προϋποθέσεις, ε, προπετούμενα μάλλον, ήταν οι συζητήσει που είχαμε εδώ στην ε, Επιτροπή μας και η συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή ότι η δουλειά αυτή που κάνουμε θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα, σε γεγονότα, προσπαθώντας να κρατήσουμε μια ισορροπία όσο γίνεται πιο συνενετικά για να έχουμε μια όσο είναι δυνατόν πιο αντικειμενική και αξιολόγηση των συνταγματικών ε, αλλαγών που έλαβαν χώρα στην Ουγγαρία και πώς επηρέασαν το δικαστικό ε, σύστημα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στα δύο πρώτα έγγραφα εργασίας μας. Το πρώτο έγγραφο αφορούσε θέματα κατάργηση εξουσιών, όπως είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που ε, συντάξαμε τον κύριο Έγγελ από το ΕΛΚ. Το δεύτερο είναι θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδη αρχές που ε, συνέταξα από κοινού με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Αγγιλάρ, και σήμερα το τρίτο έγγραφο εργασία που με χαρά συνυπογράφω με την κυρία Βέμπερ. Σύντομα θα έχουμε και ένα τέταρτο έγγραφο εργασία για θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου ώστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πάζλ, αυτό το τοπίο ε, που αφορούν την Ουγγαρία και απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αυτά εκφράστηκαν στο ψήφισμα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έγγραφο εργασία το έχετε λάβει. Εγώ είμαι κυρίως εδώ για να ακούσω κατά κύριο τα δικά σας θέματα που σας απασχολούν ή ερωτήσεις για συγκεκριμένα γεγονότα, δεδομένα που θέλετε να ρωτήσετε. Επίσης, αν θέλετε να σχολιάσετε το έγγραφο, η κυρία Βέμπερ που εργάζεται με αυτόν τον θεμάτων γενικότερα, δεν θέλω να την προκαταλάβω, θα ήθελα η ίδια να τοποθετηθεί για τα ζητήματα που μας ανησυχούν σε μια συγκεκριμένη χώρα της Ένωσης. Οπότε ελτάχει μόνο να φερθώ σε αυτό το έγγραφο, όπως είπα. Το έγγραφο αυτό είναι κομμάτι μιας ε, εργασίας ανεξελίξης, συνεργασία με τις ε, Ουγγρικές Αρχές και άλλες, ε, άλλους θεσμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν μια δουλειά που είναι σε εξέλιξη ακόμα. Αναφερόμαστε σε αυτούς τους νόμους της Ουγγαρίας που ήδη από τον Αύγουστο 2010 για σειρά νόμων παραθέτει ο μιλητής του 2010 και ήταν μεταξύ των πρώτων νόμων στην Ουγγρική νομοθεσία που επισημάναμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτέλεσαν αφορμή για συζήτηση ε, και έδωσε στην Επιτροπή και μετά στο ψήφισμα που ε, πέρασε από την Ολομέλεια αξίζει να πει κανεί ότι αυτό το ψήφισμα και τι συζητήσει ξεκίνησαν ένα διάλογο με τι Ουγγρικέ Αρχέ που έχει αποφέρει κάποια αποτελέσματα. Το έγγραφο λοιπόν εργασία μα, ε, μεταξύ άλλων προσπαθεί να δώσει μια γενική εικόνα ε, και των εξελίξεων και προς τα που κινείται ο διάλογος την εισαγωγή βλέπετε κάνουμε μια επισκόπηση των νόμων που είναι σημαντική για το θέμα μας. Έπειτα έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, την εκτίμηση που έχει κάνει ο ΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ακαδημαϊκοί φορείς, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απάντησε στα ερωτήματα και τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προέβηκε σε κάποιες διαπραγματεύσεις με τις Ουγγρικές Αρχές για κάποιες τροποποιήσεις στην Ουγγρική νομοθεσία, ιδίως σε θέματα δικαίου περιταγωνισμού, αλλά και όχι μόνο, και άλλα ζητήματα που αφορούν την αρχή της χώρας καταγωγής και όλα όσα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή αυτού του νόμου. Τώρα, ευρύτερε ανησυχίε ε, που εξέφρασε το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ε, αναφέρουμε στο κείμενό μας και θέματα που αφορούν την εξαρτησία των συντακτών του τύπου, άλλα θέματα που αφορούν της, το ευρύ πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων καταχώρησης ε, που προβλέπει ο νέος νόμος. Είναι κάτι που επεσήμανε ιδιαίτερα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η καταχώρηση κατέστη υποχρεωτική για όλα τα ΜΜΕ, όλες τις κατηγορίες, ακόμα και για όσο είναι στο διαδίκτυο. Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ευρύτερες, γενικότερες από αυτές που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, κάτι πιο σημαντικό είναι η απόφαση του ίδιου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας η απόφαση 165 του 2011 η οποία αποφάσισε τη διαγραφή κάποιων διατάξεων αυτών των νόμων ιδίως αναφέρομαι στο νόμο 104. Η απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου οδήγησε κάποιες προσαρμογές και αλλαγές ε, σε αυτούς τους προναφερθέντες νόμους. Βλέπετε λοιπόν στο εγγραφό μας προβαίνουμε σε μια περιγραφή ε, των ανταλλαγών απόψεων στις ευρωπαϊκές αρχές, την εκτίμηση που έχουν κάνει διάφοροι φορές και οργανισμοί. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος ε, του εγγράφου εργασία μας. Επίσης με αναφέρουμε τις αλλαγές που έγιναν στο μεσοδιάστημα από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και Επίση, απαριθμούν τις απαντήσεις που έδωσαν ε, διάφορες οπλικές αρχέ και η κυβέρνηση και από το σημείο 4 και μετά αναφέρουμε έναν κατάλογο των εκκρεμών α, ζητημάτων όπως απαιτήσεων καταχώρησης για τα ΜΜΕ, κάτι που περιορίζει θεωρούμε την ελευθεροτυπία, άλλες ε, ανησυχίες φορούν το περιεχόμενο τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο των ειδήσεων, τον περιορισμό της διάδοσης ειδήσεων και ε, απόψεων μέσω των ΜΜΕ και τις διαδικασίες για το διορισμό του Προέδρου του ε, Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου ε, των Μέσων Ενημέρωσης. Η διαδικασία για το διορισμό του Προέδρου σε αυτό το Συμβούλιο φαίνεται να γίνεται πολύ άμεσα, χωρίς να είναι μια ανοιχτή διαδικασία, με πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να υπάρχει και κάποιος έλεγχος. Άλλες ανησυχίες που εκφράζουμε αφορούν την ίδια τη θητεία και το κατά πόσον η θητεία πρέπει να πάβει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή όχι και τον υπάρχουν πληρωτέ ή όχι για αυτή τη θέση. Α, αυτά για αυτό το έγγραφο εργασία. Θα ήθελα πολύ να ακούσω, Μήπω πρώτα απ' θα μιλήσει και η συνεισηγήτρια, κυρία Βέμπερ, να παρουσιάσετε σε αλλά από εκεί πέρα θέλω να ακούσω και τις δικέ σα απόψει, σχόλια, επικρίσεις και πριν κλείσω ευχαριστώ θερμά τη Ρενάτα Βέμπερ για τη συνεργασία που είχα μαζί της και με το γραφείο της, όπως και την γραμματεία και ιδίως την κυρία Τσέχιου για τη βοήθεια που μας παρήχε και επαναλαμβάνει ο μιλητής ότι είναι έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. by uh, our colleagues with Tavares. Um, Μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Ταβάρες, θα ήθελα να κάνω μερικά γενικά σχόλια. Αφού συζητάμε την κατάσταση ως προς τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία και αλλού, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν το διαχωρίζουμε από την υπόλοιπη κοινωνία. Πρέπει να ξέρουμε, να βλέπουμε ολόκληρη την Ουγγρική κοινωνία και να εξετάζουμε το θέμα της ελευθεροτυπίας σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε από τα υπόλοιπα θέματα και από την υπόλοιπη πραγματικότητα της μεταρρύθμισης της Ουγγρικής Διοίκησης και Κοινωνίας. The Γι' αυτό τα νομικά κείμενα είναι το ίδιο σημαντικά με το, με το πώς τα βλέπουν οι άλλοι. Και πρέπει να πούμε λοιπόν ότι όσοι εργάζονται στην Ουγγαρία στα μέσα δεν αισθάνονται καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι. Δεν θεωρούν ότι η δημοσιογραφική τους ζωή έχει διευκολυνθεί ή ότι εκτιμάται ιδιαιτέρως ή ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Σωστό είναι βέβαια ότι κατά την επίσκεψή μας στην Βουδαπέστη είδαμε και ανθρώπους που δούλευαν εκεί σε αυτό το τομέα και με μερικές ελάχιστες εξαιρέσεις και μερικούς που συνεργάζονταν στενά με την κυβέρνηση. Όλοι αυτοί μας είπαν ότι αισθάνονται τουλάχιστον περίεργα για την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Το θέμα λοιπόν είναι τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση για να διορθώσει μια τέτοια κατάσταση ή αντίληψη. Και η σωστότερη απάντηση θα ήταν νομοθεσία και συμπεριφορά που να δίνει όσο δυνατόν περισσότερες εγγυήσει για να μπορούν όσοι εργάζονται στα μέσα να αισθάνονται προστατευμένοι ότι προστατεύεται η ελευθερία τους για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ουγγαρία. Αν και έχουν σημειωθεί μερικές αλλαγές, με βάση αιτήματα της Κομισιόν. Πάντως, πώς να το πω τώρα, οι πιο τρομακτικές διατάξεις ακόμα ισχύουν και μπορεί κάποιος διοικητικός έλεγχος που μπορεί να διαταχθεί με διάφορους τρόπους να επιφέρει τελικά κάποια πίεση στη γραμμή που θα ακολουθεί κάποιο μέσο ενημέρωσης. Ο διορισμός των δημοσιογράφων γίνεται και με κυβερνητική παρέμβαση, δεν αποκλείεται αυτό. Εξαρτάται από το πόσο θέλει η κυβέρνηση να μας πείσει ότι δεν θα παρέμβει, ότι ο τύπος είναι ανεξάρτητος, αλλά πρέπει να δοθούν και νομικές εγγυήσεις ως προς τις διαδικασίες των διορισμών κτλ. Και αυτά δεν είναι μόνο δικές μου προσωπικές ιδέες. αλλά τα ζήτησε και το Συμβούλιο της Ευρώπης ανεξάρτητοι εμπειροχνόμονες και αυτά είναι και τα συμπεράσματα του ΟΣΑ και γι' αυτό το συγκεκριμένο μου ερώτημα προς την Κομισιόν είναι τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι όλες αυτές οι συστάσεις θα εφαρμοστούν διότι από πολιτικής απόψεως καθήκον του Κοινοβουλίου μας είναι να ψηφίσει κάποιο ψήφισμα, να γράψει μια έκθεση, αλλά από πρακτικότερης απόψεως η Κομισιόν έχει τα μέσα για να συνεργαστεί με την Ουγγρική κυβέρνηση και να επιτευχθούν τέτοιες αλλαγές. Ας μην συνεχίσω γιατί τα είπε και ο κύριος Ταβάρες πριν. Θα με ενδιέφερε όμως να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι ως προς τη γενική αυτή εντύπωση που υπάρχει μεταξύ των δημοσιογράφων στην Ουγγαρία ότι υπάρχει τρομερή παρεμβολή και δυνατότητα παρεμβολής της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάντς τώρα. Σας κατευχαριστώ. Καταρχήν πρόκειται για εξαιρετική έκθεση και αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της ελευθεροτυπίας και του πλουραλισμού στην Ουγγαρία. Και επισέρχεται και σε λεπτομέρειες περί την ισχύουσα νομοθεσία εκεί εδώ και δύο χρόνια. Είναι πολύ καλή η περιγραφή των επικρίσεων που έχουν ακουστεί διεθνώς επίσης και των ανησυχιών που παραμένουν. Αυτό που δεν είδα όμως και συνδέεται και με αυτό που είπε η Ανάτα είναι τα αποτελέσματα της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάνω από δύο χρόνια δεν βλέπουμε προβλήματα μόνο στο νομικό πλαίσιο αλλά και στην επίπτωση της νομοθεσίας. Δείχνει λίγο πολύ γιατί επιμένουμε στην ανεξαρτησία των, της αρχής που είναι υπεύθυνη για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο υποκειμενικό αίσθημα αυτό. Μιλάω για τις επιπτώσεις ας πούμε πώς μιλάνε τα μέσα για τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης. Ε, τα λένε αντικειμενικά ή όχι. Υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά. Νομίζω τρεις δικαστικές αποφάσεις σχετικά που δείχνει ότι δεν δόθηκε συχνότητα σε ένα ραδιόφωνο ή δόθηκε και αφαιρέθηκε επανειλημμένος ή παραδείγματα λογοκρισίας. Μιλήσατε και για τις εκθέσεις του πρακτορείου MTI που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει μια τάση για μονοπωλιακή πληροφόρηση. το πρακτορείο αυτό τελικά οδήγησε τα υπόλοιπα σε κλείσιμο, σε πτώχευση. Και η διαφημιστική τους πολιτική επίσης οδήγησε σε στρέβλωση του όλου, της όλης κατάστασης με τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά δεν αρκεί να μιλήσουμε για το νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν και εκθέσεις που αναφέρουν συγκεκριμένες επιπτώσεις της νομοθεσίας. We, have enough. Και ίσως καλό θα ήταν επίσης σε σύνδεση και με την άλλη έκθεση που αφορά περισσότερο το πανενοσιακό πλαίσιο και συστάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για να διασφαλιστεί η ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης σε πανενοσιακό επίπεδο. Νομίζω μπορούν να συνδεθούν αυτά το νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Τι συμβαίνει στην πράξη δηλαδή αντικειμενικά, όχι μόνο υποκειμενικά. Καλό θα ήταν χρήσιμο για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταβάρης και την κυρία Βέμπερ για αυτά τα έγγραφα εργασίας γιατί έχω κάνει και εγώ τέτοια δουλειά στο παρελθόν και ξέρω τι σημαίνει. Το έγγραφο υπαριθμών 3 είναι πολύ πλήρης περιγραφή της κατάστασης αναφέρει και τις επικρίσεις και άλλα σχόλια που έχουν ακουστεί. Είναι λοιπόν και αυτό πολύτιμο για μας. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω το γενικότερο πλαίσιο. Ξέρουμε ότι η Ουγγαρία ανέλαβε μεγάλες μεταρρυθμίσεις νομοθετικές και συνταγματικές και οι αρχές ομολόγησαν ότι κατά τις αλλαγές αυτές και λόγω της φύσης τους πολλά πράγματα δεν έγιναν τέλεια. Όπως θα θέλαμε δηλαδή. Και γι' αυτό όλα αυτά δεν έχουν ακόμη τελειώσει, δεν είναι τελειωτικές οι αλλαγές. Τις επιτηρούμε, τις παρακολουθούμε, Έχουν υπάρξει και ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μας αλλά και δηλώσεις της Επιτροπής και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και κάθε φορά που κάποιο ίδρυμα έκανε βάσιμη κριτική για κάτι που έγινε στην Ουγγαρία, οι Ουγγρικές αρχές ε, το συμβάστηκαν και φαντάζομαι ότι και αυτό είναι μια διαδικασία που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτά τα έγγραφα δεν λένε τίποτα καινούριο, αναφέρουν στοιχεία ας πούμε. Φαίνεται σαν να μην ήταν ατομικό δικαίωμα η ελευθεροτυπία που το εγγυάται το Σύνταγμα, αλλά μάλλον και μόνο αποκλειστικά υποχρέωση του κράτους. Λογικό με είναι αυτό. Δεν είναι η ελευθεροτυπία το ατομικό δικαίωμα, αλλά η ελευθερία της έκφρασης. Αφού μιλήσουμε για τον τύπο, είναι λογικό το κράτος να αναλαμβάνει τη δέσμευση να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου. Πάντοτε λοιπόν μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες του τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Για τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου πράγματι εκεί έχουν ληφθεί κάτι αποφάσεις που ακύρωσαν προηγούμενες διατάξεις της Ουγγρικής νομοθεσίας όπως ακριβώς πρόσφατα έγινε κάτι ανάλογο και για τον εκλογικό νόμο. Δεν λέω με αυτό ότι ήταν τέλειος ο νόμος αυτός. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάρει την απόφαση αυτή το συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά πολλές φορές έχει υπονοηθεί ότι και το συνταγματικό δικαστήριο δεν εκφράζεται ελεύθερα και δεν δρά ελεύθερα. Έχω την εντύπωση όμως ότι το συνταγματικό δικαστήριο της Ουγγαρίας λειτουργεί καλά. Και όταν ένα συνταγματικό δικαστήριο παίρνει τέτοιες αποφάσεις, όπως και σε άλλες χώρες, αυτό δείχνει ότι δουλεύει σωστά. Και ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο μαύρα. Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό θέμα στο έγγραφο αυτό. Οι διορισμοί των εποπτικών αρχών και η σύνθεσή τους. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και στο δικαστικό τομέα, έχουν τεθεί αυτά τα προβλήματα, έχουν συζητηθεί και έχω την αντίποση ότι και αυτά είναι πράγματα που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή ότι οι Ουγγρικές αρχές έχουν συνείδηση του ότι μπορεί ο έξω κόσμος να νομίζει ότι γίνονται πολιτικοί διορισμοί για πολιτικούς λόγους και αυτό είναι μια εντύπωση που, που θέλουν να πάψει να υπάρχει αλλά τελικά νομίζω ότι οι προσπάθειές τους θα αποδώσουν. Τελικά συστήνω για να μην ακυρώσω αυτά που είπα ο ίδιος πριν από μερικούς λόγους ότι τα έγγραφα είναι αντικειμενικά αλλά απλώς φωτογραφίζουν καταστάσεις τη στιγμή που υποβάλλονται. Προβλέπεται βέβαια και μια ενδιάμεση έκθεση που φυσικά θα πάρει υπόψη της οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική εξέλιξη για να παραμείνει σε αυτή την αντικειμενική γραμμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόντς. Ε? Με συγχωρείτε που καθυστέρησα, ήμουν σε άλλη επιτροπή. Στο έγγραφο εργασίας παριθμών 3 υπάρχουν αναφορές στην προώθηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και απόψης συμφωνώ. Εδώ δεν ήρθα για να υπερασπιστώ την πρόσφατη Ουγγρική νομοθεσία. Είμαι σίγουρος ότι οι εκπρόσωποι του κυβερνώντο κόμματος θα το κάνουν καλύτερα. Θέλω όμω να πω ότι άλλες χώρες στην Ένωση μπορεί να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν αυτό το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Η Γαλλία πρόσφατα πρότεινε ένα νόμο που εγκρίθηκε που έλεγε ότι οποιοδήποτε αμφισβητεί την αρμενική γενοκτονία του 15 και την ονομάζει γενοκτονία θα διώκεται. Ε, και δεν την ονομάζει γενοκτονία. Αυτό δείχνει, ενώ η Τουρκία προβλέπει το αντίθετο, ότι και οι δύο χώρες έχουν παράλογους νόμους. Υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη όπου η έκφραση μιας άποψης που μπορεί να θεωρηθεί ως προώθηση της βίας αποτελεί αδίκημα. Υπάρχουν χώρες όπου τα πολιτικά κόμματα μπορούν να απαγορευθούν και απαγορεύονται. Πότε αυτές οι άλλες χώρες θα κατηγορηθούν επιτέλους και αυτές ή μήπω οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης αφορούν μόνο την Ουγγαρία. Κυρία Μπάλα. Ε, Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Και μη εισαγωγή να πω ότι οι όλες οι δυναμικές για την ε, νομοθεσία μετά την υιοθέτηση του νέου συντάγματος είναι κάτι πραγματικά ε, εξαιρετικό. Αν λάβουμε υπόψη ότι το Κρικό Κοινοβούλιο έπρεπε να ψηφίσει περίπου 350 νόμους, να περάσει περίπου 350 νόμους μέσα σε ένα έτος, ίσως αυτό να, αν το λάβουμε υπόψη, να εξηγεί το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι νόμοι δεν είναι απόλυτα ορθά διατυπωμένοι και περιέχουν και σφάλματα. Δηλαδή όταν ασκείται τέτοια πίεση χρονική που επέβαλε η πολιτική ηγεσία στην Ουγγαρία στον εαυτό της, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα. Πάντως, παρακαλώ, να έχετε υπόψη ότι και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο όταν ε, έχουμε πληθώρα μελετών επτώσεων να εξετάσουμε. Και αν λάβουμε υπόψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υιοθετείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, καταλήγουμε και εμείς σε σφάλματα. Έχω την αίσθηση στις λοιπόν μέσα ε, σε αυτό το πλαίσιο μπορούν ε, να υπάρξουν σφάλματα. Και ποτέ καμία νομοθεσία δεν είναι τέλεια. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω σε σχέση με τα λεγόμενα του κυρίου Έγκελ είναι ότι ευτυχώς το συνταγματικό δικαστήριο στην Ουγγαρία φαίνεται να λειτουργεί καλά και από ό,τι υπόθηκε και νωρίτερα, πρόσφατα, ε, επέκρινε το εκλογικό νόμο της χώρας και εν μέρη ε, τον κατάργησε στο δικαστήριο. Αυτό το θεωρώ ένα τεράστιο άλμα και πολύ σημαντικότερο από την ε, δράση που ανέλαβε σε σχέση με το νόμο για τα ΜΜΕ. Πολύ θετικό βήμα επίσης είναι ότι μετά από τις επικρίσεις που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και από το Σταγματικό Δικαστήριο, άλλαξε ο νόμος. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Από την άλλη, απόλυτη ελευθερία να περιμένει κανείς είναι υπερβολική προσδοκία, είναι ψευδέστηση μάλλον. Ακόμα και οι πυρογνώμονες που ήταν μαζί μας σήμερα τι μας είπαν, ότι και οι ευρωπαϊκέ αξίες ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί απόλυτα ε, σε ό,τι αφορά αξίες για την ελευθεροτυπία κάθε περίπτωση σίγουρα η Ευρωπαϊκή θα πρέπει να είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται η ελευθερία που προσδοκούμε. Πάντως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξή. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Πριν από δύο μέρες στις ειδήσει άκουσα για μια επίθεση έναντι Έλληνα δημοσιογράφου που υπερασπίστηκε τη λιτότητα που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ρωτώ τους ε, αγαπητούς συζητητές, πάντα σεβόμενοι το έργο τους. Εσείς έχετε αισθανθεί ότι υπάρχει κάποια λογοκρισία στην χώρα από την πρόσφαση που είχατε στη χώρα. Ε, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι τα ΜΜΕ επικρίνουν ισχυρά την κυβέρνηση. Για παράδειγμα στο ATV, το κανάλι ATV, μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε ε, θέλει. Μπορεί να το πει κανείς ότι είναι φιλοκυβερνητικό αυτό το κανάλι. Και πολλές άλλες περιπτώσεις. Ε, Πολλέ φορέ ο τύπος του Ουγγαρία έχει τέτοιου επικριτικούς προ την κυβέρνηση τίτλου. Ρωτώ, εσεί διαισθανθήκατε ότι υπάρχει μια κάποια λογοκρισία στη χώρα ω η τέπεια της ε, αυτού του νόμου. Και το δεύτερο μου ερώτημα απορρέει από την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που μας και νωρίτερα για την ελευθεροτυπία και τον πλουραλισμό υπήρχε νομίζω για κάποιο δελτίο τύπου νωρίτερα ε, μετά την συνάντηση με την Επίτροπο Κρούς και επεσήμαναν οι συντάκτες ότι αξιολογούν, μάλλον ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ε, της δημοσιογραφίας ε, και των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και ότι αν το κάνουν αυτό, τότε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν θα ήταν 50 αλλά 500 σελίδες. Ρωτώ λοιπόν τους ε, εξαιρετικούς εισηγητές πώς βλέπετε τα πράγματα συγκεκριμένα στην Ουγγαρία λαμβάνοντα υπόψη γενικότερα την κατάσταση. Η Ουγγαρία είναι μια ειδική περίπτωση ή υπάρχουν φαινόμενα που υπάρχουν παντού στην Ευρώπη και απλά εστιάζεται μόνο στην Ουγγαρία. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Bauer. And if Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε συνάδελφοι, επειδή και εγώ είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσωπώ την κυβερνόσα παράταξη στην Ουγγαρία, ως ε, συνάδελφος απλά να κάνω ένα σχόλιο. Όταν υιοθετήθηκε αυτό το νομοσχέδιο, για τα μέσα ενημέρωση, παρελεύει ταχύτατα η Κομισιόν ζητώντας αλλαγές. Έγιναν αυτές οι αλλαγές, τροποποιήθηκε λοιπόν το νομοσχέδιο και μετά είδαμε την απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου που εντόπισε κάποια προβλήματα σε κάποια άρθρα, οπότε και πάλι τροποποιήθηκε ο νόμος. Έπειτα Είχαμε τις αντιδράσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα και τους αρμόδιους ε, φορείς για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές τις διαπραγματεύσεις ακόμη, αλλά υπάρχουν τα κατάλληλα χέγγια και να πει κανείς ότι οι αλλαγές αυτές ακριβώς σκόπιμες θα γίνουν και είναι τα εχέγγυα, μάλλον από τη διασφάλιση που έδωσε ο ίδιος ο Ροπλωτής Πρωθυπουργός το περασμένο Σάββατο. αυτά σε ό,τι αφορά τα γεγονότα σε απάντηση του ερωτήματο κατά πόσον υπάρχει αρκετή εμπειρία για να αποτιμήσει ε, τα γεγονότα και να προβλέψει το μέλλον. Όπως είπε ο κ. Σταβάρας, είναι σημαντικό να ε, βλέπουμε τα γεγονότα. Συμφωνώ, πράγματι να δούμε τα γεγονότα και να πάμε στην Ουγγαρία, να δούμε τα να δούμε πώς δουλεύουν και να διαπιστώσετε πραγματικά ότι υπάρχει απόλυτη ελευθεροτυπία στη χώρα. Ελευθερία έκφρασης υπάρχει απόλυτα και είναι μια εμπειρία που έχετε και έχουμε όλοι και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η ελευθερία. Συναντώντας ε, ανθρώπους μπορεί να ακούσετε και κάποια παράπονα. Σκεφτείτε ίσως ότι αν δεν έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του λόγω της λιτότητας και αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται, ε, αυτό μπορεί να το εισπράξει από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα και παντού. Αυτά για τα ΜΜΕ, αλλά γενικότερα για το όλο θέμα. Όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στην Ουγγαρία αποδεικνύει ότι ναι, δουλεύει αποτελεσματικά το σταγματικό δικαστήριο. Γενικότερα τα δικαστήρια είναι εξάρτητα και κάνουν τη δουλειά τους. Και αν μετά την τελευταία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου το Γενάρη, η κυβέρνηση θα κάνει τις σχετικές αλλαγές. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει θέμα κράτους δικαίου. Στην Ουγγαρία τουλάχιστον η κατάσταση είναι πιο προβληματική από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης. Αν πάρουμε κατά μόνας και εξετάσουμε την κατάσταση σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πάντοτε κάτι θα εντοπίσουμε. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει σε ένα ερώτημα που της απευθύνθηκε. Όχι. Οπότε επιστρέφουμε στον εισηγητή. Uh, η κυρία Βέμπερ θέλει να απαντήσει σε κάποια από τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που δεν έχει σχόλια η Κομισιόν. Αυτό ήταν η πρώτη μου δήλωση. Δεύτερη. Θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία Μπάουερ. Βέβαια δεν είναι δική μου δουλειά. Να κρίνω, μπορώ βέβαια να έχω μια άποψη γιατί μια χώρα 20 χρόνια μετά την ε, μεταπολίτευση χρειάζεται να εγκρίνει πάνω από 350 νόμους μέσα σε ένα χρόνο. Στις άλλες χώρες αυτά έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 90, 90-91, γιατί τότε είχε γίνει η μεταπολίτευση όταν ιδρύεται ένα καινούριο κόμμα, έρχεται στην εξουσία μάλλον ένα καινούριο κόμμα και κάνει τέτοιες αλλαγές μπορεί να είναι ανησυχητικό το φαινόμενο γιατί δεν ξέρει κανείς, δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί. Και αναγκαστικά βέβαια αυτά τα πράγματα γίνονται βιαστικά χωρίς την απαραίτηση τη δημόσια συζήτηση. Δεν ακούγονται όλες οι απόψεις και η νέα νομοθεσία επομένως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία γενικότερα. Και υπάρχουν και αντιφατικές διατάξεις, αναγκαστικά. Δεν ξέρω αν είναι μοναδική περίπτωση η Ουγγαρία, αλλά φυσικά υπάρχουν προβλήματα για την νομοθεσία που ισχύει για τον πλουραλισμό, την ελευθεροτυπία και σε άλλες χώρες μέλη, μάλλον σε όλες αν και όχι στον ίδιο βαθμό. Στην Ουγγαρία όμως, αυτό το συζητήσαμε εξάλλου και πριν από δύο χρόνια, στις αρχές του Ιανουαρίου του 2011, στην Ουγγαρία η νομοθεσία για την ελευθεροτυπία, στην νομοθεσία αυτήν, οτιδήποτε ήταν χειρότερο από άλλες χώρες το πήραν και το έβαλαν εκεί. Και τρόμαξε ο κόσμος με την καινούργια αυτή νομοθεσία σκεφτόμενος και τις επιπτώσεις που θα είχε. Ναι, βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ελπίζω μέχρι να ολοκληρωθεί η έκθεση και να φτάσει στην ψηφοφορία να σημειωθούν αλλαγές και να χρειαστεί να την προσαρμόσουμε. Το ελπίζω αυτό. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι μετά από δύο χρόνια εφαρμογής αυτών των νόμων με μερικές αλλαγούλες, κυρίως αυτές που ζήτησε η Κομισιόν, αλλά όχι και τόσο σοβαρές. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν, ιδού οι επιπτώσεις αρχίζουν να φαίνονται. Αυτοί που συναντήσαμε στη Βουδαπέστη δεν παραπονέθηκαν για την απώλεια της δουλειάς τους για οικονομικούς λόγους. Μας είπαν ότι θεωρούν ότι πιέζονται, ότι ξαναρχίζει η λογοκρισία και αυτό είναι κάτι που μια κυβέρνηση και συμφωνώ είναι κυβερνητική υποχρέωση ο σεβασμός της ελευθεροτυπίας και επειδή ακριβώς έχει αυτή την υποχρέωση πρέπει να εγγυάται κατά 100% και παραπάνω αν γίνεται επερβάλλοντας βέβαια, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και η ίδια αρχή με τον ίδιο άνθρωπο είναι στη θέση της εδώ και δύο χρόνια. Θυμάμαι όταν συναντήσαμε εκπροσώπους του δικαστικού τομέα ότι μας είπαν ότι οι δικαστές που υποχρεώθηκαν να βγουν σε σύνταξη στα 60 δεν πρόκειται, μπορεί να επανέλθουν στη δουλειά τους αλλά ποτέ στην ίδια θέση ως προέδροι δικαστηρίων κλπ. Αυτό είναι πολύ κοινικό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για δημοκρατία βέβαια. Και φοβάμαι ότι το ίδιο γίνεται και με τους δημοσιογράφους. Πράγματι υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο που εξετίμησα ιδιαίτερα τη δουλειά του στην Ουγγαρία γενικότερα, αλλά το γεγονός είναι ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε όλοι ειλικρινά ότι γρήγορα πολλοί και από τους δικούς του δικαστές θα αναγκαστούν να παραιτηθούν. Και τότε θα δούμε αυτό το καινούργιο συνταγματικό δικαστήριο αν θα λειτουργεί γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν ακουστεί τέτοιες κατηγορίες και φήμες. Κύριε Σταβάρης. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους ε, Βέμπερ, Ούμς, Έγγελ, Μπρόνς, Μπάουερ και εσάς την ίδια, κυρία Πρόεδρε, για τα σχόλιά σας. Το modus operandi που επιλέξαμε δεν είναι το σύνηθες. Συνήθως δεν έχουμε όλα αυτά τα ε, κείμενα εργασία μαζί από τους ηγητές και τους κοιόδης. Το τρίτο εξετάστηκε, εξετάζεται, σε λίγο προβλέπεται και το τέταρτο. Και χαίρομαι γι' αυτό και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τους συνυπογράφοντες είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα και τους Ούγγρους ιδιαίτερα τουλάχιστον να σταθούν όλοι μαζί προασπίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι σημαντικό οι πολίτες να καταλάβουν ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε διαφορετικούς τρόπους εργασίας και διάφορους τρόπους εργασίας και μεθόδους και ύφος εργασίας. Πότε τα θέματα είναι πιο αμφιλεγόμενα, πότε όχι. Αλλά πάντοτε θέλουμε να κάνουμε μία αντικειμενική εξέταση το αντικείμενό μα βέβαια είναι δύσκολο αυτή τη φορά, αφορά νομοθετικέ αλλαγέ, συνταγματικέ αλλαγέ, διοικητικέ αλλαγέ. σε αυτό το συγκεκριμένο εθνικό πολιτικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο λοιπόν το θέμα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα τα περιγράψει όλα απολύτως και απολύτως αντικειμενικά. σε αυτό θα περιοριστώ ότι δηλαδή σε αυτό θα περιοριστώ επαναλαμβάνω αλλά θέλω να επαναλάβω ότι ήταν πολύ ικανοποιητικό ο τρόπος αυτός της συνεργασίας κανείς δεν μπορεί πια τώρα να πει ότι τα είδαμε πρόχειρα τα πράγματα η επιπόλαια διότι κάναμε δημαγωγική συζήτηση. Για κανένα από αυτά τα έγγραφα εργασία δεν είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Και θα προσπαθήσω να συνεχίσω να είναι έτσι τα πράγματα και στο τρίτο έγγραφο και στο τέταρτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι το έγγραφο είναι σοβαρό. Ξέραμε βέβαια από την αρχή ότι θα ήταν πολύ δύσκολο έγγραφο γιατί αφορά ένα χώρο που από τη μια είναι υποκειμενικός και από την άλλη συνεχώς αλλάζει. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκούνς ότι δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι το μισό από αυτό το περιβάλλον λείπει. Αυτό οφείλεται στο ίδιο το αντικείμενο γιατί είναι δύσκολο όπως σας είπα να το περιγράψουμε πλήρως. Αλλά επίσης οφείλεται και σε άλλους παράγοντες επιτόπου θα έπρεπε να είχαν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας που υπάρχει εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Και η ίδια η αρχή που είναι υπεύθυνη για τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να το είχε αναλάβει, η δουλειά της είναι, όπως και σε άλλες χώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να ικανοποιηθούμε με την απλή εντύπωση ότι υπάρχει πλουραλισμός, δεν υπάρχει λογοκρισία επειδή απλώς αυτά που ακούμε στο ραδιόφωνο μας φαίνονται καλά. Εδώ χρειάζεται μια ακαδημαϊκή πειθαρχία και οι εθνικές αρχές έχουν υποχρέωση να την εφαρμόζουν για να αξιολογούν τι συμβαίνει. Πρέπει να γίνουν μελέτες και έρευνες. Να υπάρξουν κοιτία παραπώνων ανώνυμα για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να μας πούν αν θεωρούν ότι υπάρχει λογοκρισία ή αυτολογοκρισία. Δύσκολα πράγματα αλλά όχι αδύνατα. Το πρόβλημα είναι ότι το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε αυτό, δεν μπορεί μέχρι τώρα τουλάχιστον να αναλάβει τέτοιες έρευνες. Μπορεί όμως σίγουρα να δηλώσει ότι έπρεπε ή πρέπει να γίνουν τέτοιες έρευνες. Το ίδιο για τον πλουραλισμό. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να οριστεί. Υπάρχουν εδώ πολιτικές, διάφορες πολιτικές ομάδες. Συμμετέσχουν όλες στη συγγραφή, ήταν πλουραλιστική η μέθοδος και το μόντους operandi αν υπάρχει μια κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή που αποτελείται από μέλη μόνο ενός κόμματος δεν πρόκειται για πλουραλισμό. Το ίδιο ισχύει για, τη... για τα μονοπόλια στις πηγές της πληροφόρησης. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν μονοπωλιακές, μονοπωλιακά πρακτορία. Αυτό φυσικά δεν είναι πλουραλιστικό. Γιατί όπως σας είπα και πριν δεν είναι και τόσο δύσκολο να ορίσουμε τι είναι πλουραλισμός. Και εδώ δεν υπάρχει. Η ομάδα υψηλού επίπεδου ευτυχώς ήρθε εδώ και πολλοί από αυτούς που έμειναν μέχρι τώρα είχαν ακούσει τι μας είπαν για το θέμα του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια το θέμα δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Τι μας είπαν λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να καθορίσουν το πλαίσιο που θα εγγυάται την ελευθερία και τον πλουραλισμό. και η Ένωση πρέπει να καθορίσει το γενικότερο πλαίσιο και να μας αναλύσει ποιες ακριβώς εγγυήσεις πρέπει να δώσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν φυσικά. Και εδώ συμφωνώ με τη Ρενάτα Βέμπερ γιατί δεν θέλησε να σχολιάσει από αυτού η Κομισιόν. Η κυρία Μπάουερ είπε υπάρχει λογοκρισία είναι και αυτό ένα ερώτημα, αλλά όχι το μόνο δηλαδή. Αν πάρουμε σοβαρά την υποχρέωση που μας δίνουν οι συνθήκες, το θέμα δεν είναι αν υπάρχει λογοκρισία, αλλά αν θα μπορούσε να υπάρξει, άμα οι νόμοι είναι γραμμένοι σωστά, θα μπορούσε να ήταν λογοκρισία ή να συνιστά λογοκρισία η σύνθεση με τον α ή β τρόπο μιας επιτροπής, αν οι εκδότες θεωρούν ότι μπορεί να κλείσει το κανάλι τους άμα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η Ένωση δεν αντιδρά μόνο εκ των υστέρων, δεν πρέπει να αντιδρά μόνο εκ των υστέρων, αλλά θέλει και να προβλέψει την ύπαρξη λογοκρισίας. Για τα δικαστήρια, ναι, τα δικαστήρια λειτουργούν διαπιστώσαμε τι αποφάσισαν και τι, πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές, αλλά ας μην το σχολιάσω γιατί υπάρχουν άλλα ή δύο έγγραφα εργασίας γι' αυτό. Τέλος, τα σχόλια Μπρόνς και της Προέδρου. Η Ένωση δεν είναι τέλεια, ποτέ δεν είχε υπάρξει τέλεια και γι' αυτόν τον λόγο ακόμη την οικοδομούμε γιατί ξέρουμε ποια είναι η προϊστορία μας ούτε αυτή ήταν τέλεια και ναι υπάρχουν πολλά προβλήματα οφείλονται πολλά στην κρίση της Ευρωζώνης ως κανονικός πολίτης απλός και αναγνώστης εφημερίδων στη χώρα μου τα βλέπω, τα διαβάζω το θέμα δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία αλλά και άλλες χώρες και ως ακαδημαϊκός θεωρώ και εγώ ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν πρέπει να παραβιάζεται. Η ακαδημαϊκή δε έρευνα να μην είναι παραπλανητική κλπ. Όλα αυτά έχουν ακουστεί ως επικρίσεις και για άλλες χώρες μέλη. Εγώ ασχολούμαι με αυτήν βέβαια. Αλλά δεν θα κάναμε καλά τη δουλειά μας αν δεν θέταμε τα προβλήματα με τον ίδιο σοβαρό τρόπο σε όλες. Αν δεν απατώμε, αυτά είχα να σας πω. Μα το εδώ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρης. Αύριο θα αρχίσουμε στις 9.30 με τους συντονιστές. Και στις 11 θα αρχίσουμε το, την τακτική συνεδρίαση. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε.